Okay, Ωραία, συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε με το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με τον Hans Hungergorst, πρόεδρο του ε, Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, τον οποίο καλωσορίζουμε θερμά στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Είναι πρώην Υπουργό Οικονομικών των Κατοχωρών και έρχεται εδώ στην Επιτροπή μας ως ε, πρόεδρος ε, ε, του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που από το 2012 ετοιμάζει διεθνή λογιστικά πρότυπα και είναι η δεύτερη φορά που τον καλωσορίζουμε εδώ με την ιδιότητά του αυτή. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ επίκαιρη ευκαιρία για να συζητήσουμε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τα λογιστικά. Στα ε, πλαίσια της ε, τρέχουσας μεταρρύθμισης ε, του ενεργολογικού πλαισίου, καθώς επίσης και λόγω των επερχόμενων νέων διατάξεων IFRS 9, 4 και οτιδήποτε άλλο έχουμε υπατμών. Ε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και η Επιτροπή μας θεωρώ ότι θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα το θέμα των λογιστικών και στο πλαίσιο της ε, νέας διακυβέρνησης ε, της ΕΦΡΑ αλλά και ε, λόγω του άμεσου διαλόγου που θέλουμε να έχουμε με το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Να καλωσορίσουμε λοιπόν και πάλι τον κύριο Χούχερβορστ και σας δίνω το λόγο για την εισαγωγική σας παρέμβαση διάρκειας 10 λεπτών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι εδώ με τον Φιλίπ Ντονζού, τον συνάδελφό μου από τη Γαλλία, για να μιλήσουμε για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και την ISB. Πιστεύω ότι ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο σημαντικό να έχουμε ποιοτικέ μεθόδους στην Ευρώπη για τους λογαριασμούς, διότι με την οικονομική κρίση συνειδητοποίησαν πόσο πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τη χρηματοδότηση μέσω τραπεζών. Και γι' αυτό θέλει να δημιουργήσει μια ε, ένωση κεφαλαίου ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στην οποία θα υπάρξει καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τι επιχειρήσει. Πιστεύω ότι ε, οι μπορούν να βοηθήσουν να δώσουν οξυγόνο ε, και κεφάλαιο στις νέες επιχειρήσεις. Ε, για να λειτουργήσουν ε, όμως αισίως αυτές οι κεφαλαιαγορές θα πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα όταν λειτουργούμε βραχυπρόθεσμα και υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων δεν λειτουργούν σωστά οι αγορές και χρειάζεται ρύθμιση για να αποφύγουμε τις καταχρήσεις για τον ηθικό κίνδυνο όταν κάποιοι επενδύουν τα λεφτά άλλων. Ε, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι λοιπόν ε, και οι λογαριασμοί σε αυτές τις αγορές ε, οι αξιόπιστες οικονομικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για να υπάρχει εμπιστοσύνη στην οικονομία της αγοράς η ISB αυτό που επιδιώκει να κάνει είναι να, ε, υπάρχουν, να είναι υπόλογοι στην κεφαλαία αγορά και να υπάρχει διαφάνεια. Θα πρέπει να ε, φροντίσουμε εμείς ώστε να υπάρχουν αληθή στοιχεία και έχουμε δώσει πολύ σκληρές μάχες στο παρελθόν για να ε, φέρουμε στο φως του ήλιου και της διαφάνειας τα κρυφά υποκείμενα στοιχεία. Ξέρουμε λοιπόν τώρα ποιο είναι το πρόβλημα πρόβλημα με τα ε, παθητικά στοιχεία ε, ως προς ε, τις συντάξεις. Ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ποιο χρέος εκρύβεται πίσω από τις μισθώσεις αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν συνέβαινε ε, στο παρελθόν και ε, ε, έχουν υπάρξει οξύες διαμαρτυρίες από πλευράς κάποιων επιχειρήσεων κατά των προτύπων μας. Εμείς επιβάλλουμε μια πάρα πολύ αυστηρή πειθαρχία στις αγορές, πολύ αυστηρότερη σε σχέση με τους λογαριασμούς σε κρατικό επίπεδο, σε πολλά κράτη-μέλη, όπου παραδείγματος χάρη τα στοιχεία παθητικού στις συντάξεις παραμένουν και καλυμμένα. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τώρα τη, το, τα διεθνή πρότυπα και την εφαρμογή, τους, ε, την εφαρμογή των IFRS στην Ευρώπη. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ατέλειες. Δεν ισχυριζόμαστε κάτι ότι είναι, λειτουργεί τέλεια το σύστημα. Πάντως θεωρούμε ότι γενικότερα μπορεί κανείς να μιλήσει για θετικό αντίκτυπο των IFRS ε, στην Ευρώπη και θα ήθελα να εξηγήσω για ποιο λόγο είμαι τόσο αισιόδοξο. Πρώτον, θα έφερες ε, το 2005 ε, έδωσε μια κοινή λογιστική γλώσσα στην Ευρώπη και πριν από την έγκρισή τους η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια μυριάδα ε, λογιστικών γλωσσών, πάνω από 50. Συνταξιωτικά ταμεία και άλλοι θεσμικοί επενδυτές λοιπόν έπρεπε κατά το δοκούν να επιλέξουν ότι την γλώσσα τους, υπό τη λογιστική γλώσσα που θα χρησιμοποιούσαν και δεν υπήρχε μετάφραση από τη μία στην άλλη. Άλλαξαν οι κανόνες του παιχνιδιού ως προς την προστασία των καταναλωτών με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, διότι δημιουργήθηκε μεγαλύτερη διαφάνεια και εξοπιστία προς όφελος των επενδυτών και τώρα οι ρυθμιστές ε, που τώρα έχουν συγκεντρωθεί στην ΕΣΜΑ μπορούν να συγκρίνουν τους λογαριασμούς και να ε, επιβάλλουν ε, διακλαδική εφαρμογή των νομοθετημάτων. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις, όχι μόνο για τους θεσμικούς επενδυτές. Τώρα ισχύουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και η ικανότητα δυνατότητα να λειτουργούμε με μία μοναδική λογιστική γλώσσα σε ολόκληρη την Ευρώπη επίσης εξοικονομεί μεγάλο, ε, ε, πάρα πολλά χρήματα και για τις ίδιες εκεί για τις επιχειρήσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο ακολουθήθηκαν τα Σε 114 χώρες στον κόσμο έχουν εγκρίνει αυτά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και 12 επιτρέπουν τη χρήση. Σε ολόκληρη η Ευρώπη, ολόκληρη η Λατινική Αμερική, Καναδά, οι περισσότερε ασιατικές χώρες, όλες χρησιμοποιούν ε, διεθνή λογιστικά πρότυπα και το ίδιο ε, ευρύως διαδεδομένη χρήση του σε επιχειρήσεις της Κίνας και της Ιαπωνίας. Ε, αντιστέκονται οι ΙΠΑ, αλλά ακόμη και εκεί οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν στα χρηματιστήρια, τα IFRS για τις εισηγμένες στα εκεί χρηματιστήρια ε, ε, εταιρείε. Ε, η διάδοση των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι πάρα πολύ μεγάλο όφελος για θεσμικούς επενδυτές όπως τα συνδεξιδετικά ταμεία. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές ώστε να έχουν καλά, καλές απολαβές, καλά αποτελέσματα για τους ε, συνταξιούχους ε, και το ίδιο ισχύει για πολλές κορεατικές, ε, βραζιλιάνικες επιχειρήσεις παραδείγματος χάρη. Έχει μειωθεί το κόστος, έχει μειωθεί το κόστος του κεφαλαίου και το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις θηγατρικές εταιρείες. Η συντριπτική πλειοψηφία των 114 χωρών που έχουν εγκρίνει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα το έχουν κάνει χωρίς να χρειαστούν τοπικές προσαρμογές. Το ότι δεν έχουν το ότι δεν έχουν διαμαρτυρηθεί κατά των προτείνων δεν σημαίνει ότι συμφωνούν με όλα αυτά που λέμε. Πάντως, εάν αρχίσουν όλοι να πειράζουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και να κάνουν προσαρμογές, τότε θα εξανεμιστεί το όφελος των διεθνών λογιστικών προτύπων και θα επανεθνικοποιηθούν τα πρότυπα. Ε, πέρα από κάποιες λιγοστές εξαιρέσεις, μπορούμε να πούμε ότι η Ευρώπη έχει υιοθετήσει τα λογιστικά πρότυπα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χωρίσει την κυριαρχία τη ω προ τα λογιστικά πρότυπα η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρώπη δεν ε, δέχεται ασυζητητή τα πρότυπά μας ε, και ε, ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει μια από τις πιο περίπλοκες διαδικασίες έγκρισης. Υπάρχει ο ΙΦΡΑ και υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο που πρέπει να εγκρίνουν τα πρότυπα και εμείς στην ISP ξέρουμε ότι εάν δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη την άποψη Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε θέτουμε εν κινδύνο την έγκριση των λογιστικών προτύπων. Δεν σας θεωρούμε δεδομένους χοντρικά. Το αντίθετο ταυτόχρονα ελπίζουμε ότι η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι ως διεθνής οργανισμός δεν μπορούμε να μας επιτρέψουμε να ακούμε μόνο ε, τους ευρωπαϊκούς ε, οργανισμούς. Θα πρέπει να ε, εισακούμε τις επιθυμίες όλων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, προσπαθούμε βάσει των παρατηρήσεων σας όταν το κρίνουμε σκόπιμο να λάβουμε υπόψη τα σχόλια σας. Ε, ξέρουμε ότι οι οικονομικές δηλώσεις παραδείγματος χάρη παρά είναι ε, μεγάλες και αναθερούμε τώρα τα πρότυπα μας για τις αποκαλύψεις στοιχείων. Υπάρχουν ε, κάποιοι επενδυτές ε, επίσης ε, που φοβούνται ότι δεν ευσταθούν οι αποτιμήσεις που γίνονται, οπότε θα προτείνουμε προληπτική εποπτεία ούτως ώστε να μην υπερτιμάται η αξία των ενεργητικών και να μην υποτιμάται η αξία των στοιχείων του παθητικού Χρειαζόμαστε όμως ανεξαρτησία για να αποφύγουμε τα ίδια συμφέροντα όπως και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών πρέπει να είναι ανεξάρτητοι ως προς την πολιτική ζωή και τις επιχειρήσεις. Ε, πάντως το ρυθμιστικό κομμάτι είναι σημαντικό αντίβαρο για την οικονομική κρίση. Θα σας ακούσουμε όλους αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπερασπιστούμε το δημόσιο συμφέρον. Ας καταλήξω και σε κάποια συμπεράσματα κυρίες και κύριοι. Καλωσορίζουμε τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει μια ένωση κέφαλαια αγορών η ε, χρήση ε, νέου συστήματος προτύπων όπως τα διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι ε, εκ των όνου κάνεφε για να λειτουργήσουν σωστά οι κεφαλαίοι Μόνο με σωστή ρύθμιση μπορούν να λειτουργήσουν εύρυθμα και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της νομοθετικής ρύθμισης και η ISP θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πετούμενα εργαλεία για να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες Σα Ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε μας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εισαγωγή σας. Και τώρα θα δώσω αμέσω τον λόγο στους αγορητές. Ο πρώτος ο κύριος Μπάλτς παρακαλώ. Ευχαριστώ θερμά πρόεδρε. Η, ε, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εργάζεται με βάση και τις ε, ε, δυνατότητες για τις ε, διαφορετικές πράξεις και για τις δυνατότητες αντανάκλασης των οικονομικών στοιχείων. Πώς μπορούν οι, τα δύο διαφορετικά αυτά πρότυπα να είναι συνεκτικά μαζί τους και πώς μακροπρόθεσμα όσον αφορά τις ασφαλίσεις μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη τους. Δεύτερη ερώτηση ως ε, ε, περαιτέρω εναρμονιστική δυνατότητα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την προσέγγιση με κριτικό πνεύμα να φωτίσω το τι γίνεται και την λειτουργικότητα να δούμε τι συνεπάγεται για τη λειτουργικότητα. Δεν μπορεί να είναι προ όφελο ε, ε, του θεματολογίου της ανάπτυξης όσον αφορά τις μικρομεσές επιχειρήσεις που θα πρέπει να χρηματοδοτούνται οι διεθνείς ε, προδιαγραφές και τα διεθνή πρότυπα και να μην λαμβάνονται υπόψη οι αναλύσεις κόστους. Και μακροπρόθεσμα ήδη εδώ βρισκόμαστε ίσως μπροστά σε ένα νέο εναρμονισμό. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ολοκληρώσει από πλευράς μας και βρισκόμαστε στην διαδικασία εργασίας ε, όσον αφορά την ε, ε, δυνατότητα προδιαγραφών επί της ουσίας και πολιτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο δυσχερές εγχείρημα και πολύ σημαντικό για τις βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Πολύ σωστό αυτό. Δεν έχουμε ακόμα δρομολογήσει Πρέπει ακόμα να ολοκληρώσουμε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα όσον αφορά. Δεν έχουμε ακόμα τις ε, τελικές ημερομηνίες και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την διάδραση που υπάρχει και να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις. Αλλά δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει τις αντιστοιχίες λογιστικά και μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ο καλύτερος τρόπος μακροπρόθεσμων επενδύσεων είναι να αγοράζουν ομόλογα και μετοχές ε, οι ενδιαφερόμενοι και αυτό υπάρχει, ε, εν ε, υπάρχουν κίνδυνοι σε αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επενδυτές να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στις ε, συμβουλές και όσον αφορά τις εταιρείε, ώστε να έχουν μια σωστή εικόνα του τι συμβαίνει. Περί αυτών έχουμε ιδιαίτερη σπουδαιότητα για αυτές τις λογιστικές πρακτικές και τα λογιστικά πρότυπα, για τις ευκαιρίες που προσφέρουν, αλλά επίσης και τους κινδύνους που μπορεί να αξιολογήσει μια εταιρεία με βάση αυτά αυτά τα στοιχεία. Είναι τεράστια σπουδαιότητα να έχουμε όλε αυτέ τι πληροφορίε σε σχέση με του ισολογισμού ώστε να αντανακλώνται και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Καθώς αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μια μικρομεσαία επιχείρηση αν δεν είναι καταχωρημένη, αν δεν έχει εγγραφεί σε ένα χρηματιστήριο, είναι ιδιαίτερα περίπλοκες οι προδιαγραφές και οι διατάξεις για αυτήν. Είναι απόφαση όμως όχι δική μας. Είναι οι ρυθμιστές ε, των ε, ε, θεμάτων ασφάλισης που πρέπει να ευθυγραμμίζονται όλες οι καταχωρημένες σε χρηματιστήρια εταιρείες όσον αφορά τις μεγαλύτερες αλλά και κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη μεγάλη τους πλειοψηφία όταν είναι μια καταχωρημένη εταιρεία σε ένα τέτοιο χρηματιστήριο πρέπει να ευθυγραμμίζεται με αυτές τις αρχές ώστε οι επενδυτές να μπορούν να βασίζονται σε αυτά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Είναι όμως ε, οι ρυθμιστές όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας οι υπεύθυνοι για αυτά. Αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε σε σχέση με το σύστημά μας είναι να μειώσουμε τον περίπλοκο και ιδιαίτερα σύνθετο χαρακτήρα αυτών των στοιχείων. Προσπαθούμε να απλουστεύσουμε με τέτοιο τρόπο την λειτουργία τους ώστε οι εταιρείε να το θεωρούν και να μπορούν να το χρησιμοποιούν ευκολότερα για να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Τώρα για τους σοσιαλδημοκράτες ο κύριος Μπαγιέ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξέρω καταρχάς ε, με όλα όσα έχουμε αυτή τη στιγμή στα IFRS e ποια είναι τα συγκεκριμένα σχέδια τα οποία έχετε σε κάποιες χώρες, θεωρείτε ότι μπορούν να υλοποιηθούν αυτά και αν έχετε κάποια σχέδια για να μπορέσετε να υλοποιήσετε κάποια πράγματα. Και επίσης είπατε ότι οι επενδυτές σίγουρα θα πρέπει να ε, έχουν εμπιστοσύνη στους κινδύνους που πρέπει να αναλάβουν. Αυτό ισχύει βέβαια και για το ε, για την κοινή γνώμη και για διάφορες χώρες και στο Βέλγιο και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης ε, και αμφισβητείται λίγο όχι τόσο η εφαρμογή του κανόνα SA 2010 αλλά με την εφαρμογή αυτού του διεθνούς κανόνα ουσιαστικά υποχρεώνουμε τις ε, δημόσιες αρχές να ε, υπολογίζουν σε ένα χρόνο και να κάνουν ε, λογιστικό ε, υπολογισμό ε, τα πάντα και εμείς δεν μπορούμε να δούμε έτσι τι αποθεματικό μπορεί να έχουν οι δήμοι, οι κοινότητες ή και μια ολοκληροχώρα χώρα. Εξετάζεται το θέμα αυτό. Ξέρω ότι η συνθήκη προβλέπει να χρησιμοποιούμε και να αναλύουμε μόνο τις ε, δαπάνες και το χρέος, αλλά κάπου θα πρέπει ε, να δούμε και ότι το συνολικό χρέος δεν είναι το καθαρό χρέος, είναι και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούμε να έχουμε ως ε, κληρονομιά και να μπορούμε να συνυπολογίσουμε και αυτά. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν την άποψή σας επ' αυτό. Ναι. Ο συνάδελφος θα μπορέσει να σας απαντήσει στο δεύτερο ερώτημα στα γαλλικά. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα τώρα που αντιμετωπίζουν όλοι όσοι παγκοσμίω εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ε, Συνήθω έχουμε διαμαρτυρίε ε, ω προ την πολυπλοκότητά του και αν το εξετάσουμε αυτό, η πολυπλοκότητα προέρχεται από περίπλοκες ε, επιχειρηματικές δραστηριότητε. Πολλές ε, επιχειρήσεις έχουν ε, προβλήματα με, την, ε, ε, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και υπάρχει παθητικό εκεί. Υπάρχουν επίσης θέματα χρηματοοικονομικών παραγόγων, εκεί περιπλέκονται περισσότερο τα πράγματα. Αλλά για επιχειρήσεις που σχετικά, έχουν σχετικά απλά επιχειρηματικά μοντέλα, το IFRS δεν είναι και τόσο δύσκολο. Και το εκπληκτικό είναι ότι αν δείτε ότι 114 χώρες παγκοσμίως έχουν ε, υιοθετήσει τα πρότυπα αυτά και ε, πολλά ε, από αυτά τα κράτη δεν έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα και αναδυόμενες χώρες όπως η Βραζιλία, η Κορέα, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη βέβαια ούτως ή άλλως είναι ήδη ανεπτυγμένη, αλλά οι χώρες αυτές καταφέρουν να εγκρίνουν τα διεθνή πρότυπα χωρίς πολύ σοβαρά προβλήματα. πρόσφατα μίλησα και με επιχειρήσεις εσωτερικών ελεκτών ε, για τις εντυπώσεις που έχουν ε, και ε, για την εφαρμογή σε αυτές τις χώρες και λένε ότι είναι πολύ ψηλό το ποσοστό εφαρμογή είναι σχεδόν συγκρίσιμο με την Ευρώπη. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, αν κατάλαβα καλά, που εξετάζει τι γίνεται και με, με τα μη λογιστικά στοιχεία και πώς προσμετρώνται αυτά στο δημόσιο χώρο, χρέος, να σας πω ότι το δημόσιο χρέος είναι καθαρά εκτός αρμοδιότητας του δικού μας του οργανισμού. δεν τα εκπονούμε εμείς τα πρότυπα για τις ε, κοινότητες, τους δήμους κλπ. Υπάρχει ε, άλλος οργανισμός ε, πυρογνωμόνων σε λογιστικά στοιχεία αυτής της μορφής το Διοικητικό Συμβούλιο του Ήψες προσπαθεί να εμπνευστεί από τους κανόνες του ε, ιδιωτικού κλάδου. Ε, έχει κάποια στοιχεία τα οποία μπορούμε να πάρουμε, αλλά φυσικά είναι διαφορετική η όλη διαδικασία. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να έχουμε τις επενδύσεις και να τις προσμετρούμε σε κάποια οικονομική διάρκεια και όχι μόνο σε ένα οικονομικό έτος. Ε, οι χώρες ε, ακολουθούν ή δεν ακολουθούν τους κανόνες ΑΕΠΣΑΣ. Κάποιες χώρες δεν υπάρχει υποχρέωση, επομένως κάποιες χώρες θεωρούν ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν. Υπάρχουν θέματα εσόδων και δαπανών και ε, λογιστικών στοιχείων ως προς τον προπολογισμό, αλλά εμείς δεν μπορούμε να εκφράσουμε άποψη από αυτού γιατί δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Ευχαριστώ. η συντονίστρια των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, κυρία Βίμπορ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση για μένα που οι Ηνωμένε Πολιτείε χρησιμοποιούν άλλο πρότυπο και όχι το IFRS και είναι και ο, ε, ακριβώς αυτός ο οποίος ε, ε, επιλέγει τελείως διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των λογιστικών θεμάτων ένα μέλος της ε, Task Force ε, για το FSB έκανε μια δήλωση στους Financial Times και είπε ότι θα πρέπει να πάνε οι τράπεζες πέρα από το IFRS 9 και να αποκαλύψουν τι απώλειες έχουν κάθε χρόνο σε σχέση με το ποσοστό που ανέμεναν και να εξηγούν γιατί υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο στοιχεία, αν τυχόν υπάρχει. Ε, αναφερθήκατε στην ολοκλήρωση της αναθεώρησης του IFRS 9. Θεωρείτε ότι ε, θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο ε, και αν όχι θεωρείτε ότι θα πρέπει να επεκταθούμε στο μέλλον στα IFRS 9 για να έχουμε ε, και κατάλληλη επιχειρηματική διακυβέρνηση εδώ. Πρώτα απ' όλα για ένα σύντομο σχόλιο για τη ΣΥΠΑ. Είναι απογοητευτικό ότι δεν έχουν ενταχθεί ακόμα σε αυτή την προσπάθεια. Ας δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι πολύ μεγάλη η χώρα, η μεγαλύτερη κεφαλαϊκή αγορά και έχουν πολύ μεγάλη παράδοση. Είναι λοιπόν δύσκολη η κατάσταση σε σχέση με εκείνους τώρα. Αυτό που ακόμα ελπίζω ότι μπορεί να γίνει είναι ότι ίσως οι θα μπορούσαν να λάβουν μια παρόμοια απόφαση όπως η Ιαπωνία να επιτρέψουν δηλαδή ατομικά εταιρείε που βρίσκονται έναντι εταιριών των λογιστικών αυτών προτύπων να υιοθετήσουν τέτοια πρότυπα. Αυτό μπορεί να είναι μια δυνατότητα. Αυτό όμως θα το δούμε στο μέλλον. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε. Εγώ είμαι μέλος του ε, Συμβουλίου ε, Σταθερότητας ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα. Έχουμε ήδη επαφέ και έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Η δημοσιοποίηση πέρα και πάνω από αυτά τα οποία απαιτούνται όσον αφορά τα λογιστικά πρότυπα ακριβώς, πράγματι πιστεύω ότι η αποκάλυψη και δημοσιοποίηση των κινδύνων και πώς εξελίσσονται αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις δηλώσεις τους ε, ώστε τέτοιου είδους απαιτήσει, ε, παρόμοιες απαιτήσει να λαμβάνονται υπόψη. Όμως προφανώς πρώτα απ' όλα ήδη λειτουργούμε με βάση πολλές επικρίσεις ότι οι απαιτήσει δημοσιοποίησης και αποκαλύψεων στοιχείων είναι πάρα πολύ ε, επιβαρυντικές, δηλαδή επιβαρύνουν πολύ τις διαδικασίες και το έργο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και συνετοί κρίνοντας το τι ακριβώς απαιτείται. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ να δραχθώ τη ευκαιρία, ώστε ε, στην μητρική του γλώσσα να θέσω ερωτήσεις ε, προς τον κύριο Χόχερφόστ στα Ολλανδικά. Θα ήθελα να μου πείτε για τις προδιαγραφές και τα πρότυπα. Είναι σαφής ε, για τις ε, τράπεζες που για παράδειγμα πέρυσι έγινε μια ε, εξεταστική τέτοια δράση και είδαμε ότι διαφορετικά πρότυπα εφαρμόζονται από πλευράς ε, των τραπεζών όσον αφορά τις, τα δάνεια, πιστώσεις και τα παράγωγα. Και αυτό δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις για τη συγκρισιμότητα των ισολογισμών τραπεζών. Θεωρείται από πλευρά του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ότι κάτι θα έπρεπε να γίνει για να υπάρχει συγκρισιμότητα και μετά επιβάρυνση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, και θα πρέπει να υπάρχουν παρόμοιες συγκρίσιμες ε, ε, προδιαγραφές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε βάση ένα απλουστευμένο σύστημα αν θα ήταν δυνατόν. Είναι δυνατόν λοιπόν σε σχέση με αυτή την οδηγία στα διάφορα κράτη-μέλη να προχωρήσει αυτό. Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες για να γίνει κάτι τέτοιο. Να έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μια πλουστευμένη μια πλουστευμένη διαδικασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Will... Απάντηση. Ο συνάδελφός μου θα λάβει τον, την, τον λόγο για να απαντήσει μετά. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το πρώτο τμήμα της ερώτησής σας, πρώτα απ' όλα, γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά για να μπορέσουν αυτά να φωτιστούν ως προβλήματα. Κατά το παρελθόν, όπως είπα στην εισαγωγική μου παρατήρηση, δεν υπήρχε κάποιος τρόπος οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να μπορούν να συγκρίνουν τα στοιχεία των διαφόρων ισολογισμών, γιατί ήταν διαφορετικές οι γλώσσες και οι προδιαγράφες ε, ε, για τη σύνταξη τους. Τώρα έχουμε ένα κοινό παρονόμαστη. Μπορούν έτσι τα προβλήματα να φωτιστούν και να διαφωτιστούν καλύτερα. Είναι δυνατόν για τους τους ρυθμιστές, τις ρυθμιστικές αρχές να εφαρμόζονται αυτά και να επιβάλλεται η ε, συμμόρφωση με αυτές τις αρχές. Δική τους δουλειά είναι οι προδιαγραφές αυτές να τηρούνται σωστά και να, να συμμορφώνονται οι, αρμο, οι εμπλεκόμενοι με αυτές τις προδιαγραφές. Πολύ δουλειά απομένει να γίνει, έχει γίνει ήδη πολλή δουλειά αλλά απομένει και πολύ ακόμα δουλειά να γίνει. Εργαζόμαστε πολύ στενά, συνεργαζόμαστε με την ΕΣΜΑ, αν έχουν την εντύπωση ότι υπάρχουν πολλές διακυμάνσεις, μπορούν να προστρέχουν σε εμά ώστε για την προσαρμογή αυτών των ε, ε, προτύπων εμείς πάντα γραζόμαστε και παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή και σε σχέση με τις προτάσεις που μας γίνονται υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής των προτύπων μας. Απαιτείται πολύ στενή συνεργασία μεταξύ ASB και ΕΣΜΑ και αυτό ακριβώς είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και έχουμε ένα μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ αυτών των δύο οργάνων και έχουμε πολύ συχνές επαφές. Ευχαριστώ. Uh, Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα λογιστικά για το πρώτο από πλευρά ε, της δικής μας εμπλοκής δεν εμπλεκόμαστε εμεί σε σχέση με αυτέ τι προδιαγραφέ, είναι θέμα τη επιτροπή και εμεί συμμετέχουμε σε αυτές τις διαργασίε. έχουμε όμως εκπονήσει πρότυπα και προδιαγραφές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτές οι προδιαγραφές είναι διαθέσιμες από το 2009 και εδώ θα πρέπει να δούμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν έχει όμως υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι διαθέσιμος μέσω αυτό ως εργαλείο, αλλά δεν έχει επιβληθεί. Κάποια κράτη-μέλη αποφάσισαν να χρησιμοποιούν ε, για κάποιες κατηγορίες εταιριών στη δική τους νομοθεσία αυτού του είδους τα πρότυπα όμως τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται εκ των ενόντων ή για, με περιορισμένο χρόνο ορίζοντα. Χρειάζονται όμως ε, και οι, ανα, οι αναγκαίες χρηματοοικονομικές δυνατότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δούμε πώς μπορούν να χρηματοδοτούνται αυτές οι ανάγκες από τους ε, ε διαθέτοντες τα κεφάλαια και πρέπει να δούμε δεν είναι μόνο το θέμα μιας χώρας αλλά και του υπόλοιπου ε, των χωρών της ε, Ευρώπης. Και αν επρόκειτο ή πρόκειται να υιοθετηθεί αυτό θα πρέπει να μπορέσει να διασφαλιστεί αυτού του είδους ε, η συνεννόηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτού του είδους οι επαφές ώστε να μπορούν αυτά τα κεφάλαια να διασφαλίζονται και να διατίθενται όπως απαιτείται. Θα ήταν χρήσιμο ίσως αυτό. Ευχαριστούμε. Για την ενωτική αριστερά, εσείς κύριε Βεγγάς παρακαλώ. Ε, ε, Εμείς από τον πόλεμο και μετά μέχρι σήμερα ε, γνωρίσαμε πολλές αλλαγές. Έχουμε ένα καπιταλιστικό, μονοπωλιακό σύστημα πλέον. Είναι πελώρη η εξουσία των μεγάλων μονοπωλίων. Σε αυτό το πλαίσιο οι ρυθμιστικές αρχές ε, έχουν ε, έναν ενισχυμένο και σημαντικότατο ρόλο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης βρίσκονται στο κέντρο σημαντικότατων συζητήσεων. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να υποβάλω και εγώ κάποια ερωτήματα σε σχέση με την ESB και το θέμα της διακυβέρνησης εξυπακούεται ότι είναι πελώρια σημασία οι αποφάσεις ε, που λαμβάνετε εσείς ε, και επηρεάζονται δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεων. Οι μετρικές πληροφορίες που προκύπτουν είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα πρέπει να διευθετήσουμε. Ε, Ε, θα ήθελα λοιπόν ε, να σχολιάσω το ζήτημα της δημοκρατικής διακυβέρνησης ε, και της ανεξαρτησίας της ESB. Από το 2008 και μετά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δημόσιας χρηματοδότησης, πέρα από την ιδιωτική χρηματοδότηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς ακριβώς λειτουργεί ο οργανισμός σας. Επίσης, στο Συμβούλιο σας εκπροσωπούνται μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, οι μεγάλες τέσσερις όπως ονομάζονται και ξέρουμε ότι πολλά από τα μέλη του διοικητικού σας συμβουλίου προέρχονται από τέτοιες μεγάλες επιχειρήσεις. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κατοχυρώνεται λοιπόν η ανεξαρτησία σας. Ε, η σημερινή συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική και καλύπτει διάφορους τομείς δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και βλέπουμε πώς εσείς ε, ε, εκπονείτε τα πρότυπα και ταυτόχρονα ελέγχετε ε, είναι πολύ σημαντικές και οι δύο λειτουργίες ε, και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διαχωρίζονται σαφώς αυτοί οι δύο ρόλοι. Θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσετε αν θέλετε σε αυτές τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την ε, δημοκρατική λειτουργία και την ανεξαρτησία του οργανισμού σας. Ε, απάντηση. Δίκαια, δίκαια τα ερωτήματά σας και πολύ υποβάλλετε ερωτήματα για τη διακυβέρνηση και συμφωνώ πλήρως. Θα έλεγα λοιπόν ότι το Εποπτικό Συμβούλιο, ένας δημόσιος οργανισμός ε, που αποτελείται από ελεκτικές αρχές, είναι το ανώτατο όριο και το ανώτατο συμβούλιο διορίζει ε, τους ε, τα μέλη του Συμβουλίου μας. Οι εντολοδόχοι λοιπόν αληθεύει ότι έχουν εργαστεί σε κάποιες επιχειρήσεις όμως άλλοι εργάζονταν, παραδείγματο χάρη, στον Γαλλικό Οργανισμό Ελέγχου των Χρηματαγορών. Ε, ε, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ανώτερο ε, επίπεδο, εποπτικό επίπεδο που διορίζει τους εντολοδόχους και εποπτεύει την ε, λειτουργία του οργανισμού μας. Τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης είναι από δημόσιες ε, πηγές, από κυβερνήσεις, ε, από ρυθμιστικές αρχές για τις κινητές αξίες και η κατανομή γίνεται βάσει του ΑΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει ένα από τα μεγαλύτερα ποσά στον προπολογισμό του, του οργανισμού μας. Η πλειοψηφία των κονδυλίων λοιπόν είναι δημόσιας προέλευσης και ε, επιδιώκουμε να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το κομμάτι της δημόσιας χρηματοδότησης. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι ανεξάρτητοι, δεν έχουν ε, καμία σχέση με εμπορικές ε, εταιρείες, είναι πλήρη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ σε εθνικό επίπεδο αυτοί που εκπονούν τα πρότυπα ορισμένες φορές ε, έχουν εποπτικό ρόλο ή συμβουλευτικό ρόλο σε επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει όμως στην περίπτωσή μας. Εμείς απαιτούμε από τα μέλη του Συμβουλίου μας ε, να είναι απολύτως αμερόληπτοι και ανεξάρτητοι. Πιστεύω δε ότι η διαδικασία ε, είναι διαφανέστερη σε σχέση με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ε, στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι δημόσια συνεδριά, αναμεταδίδονται στο διαδίκτυο. Μπορούν ε, όλοι όσοι θέλουν να τις παρακολουθήσουν. Όλα τα έγγραφα που προκύπτουν από το Συμβούλιο είναι δημόσια. τα μέλη του Συμβουλίου απαγορεύεται να συσκέπτονται μεταξύ τους ε, όταν παρευρίσκονται πάνω από πέντε μέλη για να μην προμαγειρεύουν, αν θέλετε, τα όσα διαμείβονται συνέχεια στις δημόσιες συνεδριάσεις. Όλες αυτές οι δικλίδες ε, ε, ε εγγυώνται την ανεξαρτησία του οργανισμού μας κατά τη θέσπιση των διεθνών προτύπων. Ξαναλέω ότι υπάρχει ένα δημόσιο όργανο που εποπτεύει και εμείς θεωρούμε ότι είμαστε δημόσιος φορέας και σας είπα ότι εξυπηρετούμε αποκλειστικά και μόνο το δημόσιο συμφέρον. Σας ευχαριστώ. Ο Σβέν Γκίγκολτ από τους Πράσινους. Θα ήθελα να συνεχίσω την όλη συζήτηση, στην αρχή αναφερθήκατε στην αρχή της ανεξαρτησίας και συγκρίνατε τα καθήκοντά σας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρά το γεγονός ότι δέχομαι ότι οι κεντρικές τράπεζες ε, δικαίως ε, πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητες, διότι είναι πολύ μεγάλο το δέλεαρ από τις κυβερνήσεις ε, να χρηματοδοτούνται με τα χρήματα των κεντρικών τραπεζών. Για τον καθορισμό των λογιστικών προτύπων ε, σε πολιτική, ε, στην πολιτική επιστήμη δεν βλέπω κάποιο βάσιμο λόγο για το ειδικό καθεστώς το οποίο λαμβάνετε εσείς παραδοσιακά. Αναπτύχθηκε συν το χρόνο, συνήθως τα καθήκοντά σας ε, θα πρέπει να είναι σε διεθνείς δημόσιους οργανισμούς και σε αυτό το πλαίσιο ασχολείστε με ε, το πολύ σημαντικό ε, στοιχείο της παγκοσμιοποίησης των προτύπων. Αλλά δεν είναι λογικό για μια συγκεκριμένη περιφέρεια όπως την Ευρώπη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία προέρχονται από την Ευρώπη να μην εκλέγονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή άλλους δημοκρατικούς οργανισμούς. Δέχομαι το γεγονό ότι η Κίνα που δεν είναι δημοκρατία δεν μπορεί να εκπροσωπείται από δημοκρατικά ε, ρετό άτομο. Αλλά οι Ευρωπαίοι οι ε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να εκλέγονται με δημοκρατικό τρόπο. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πότε θα προτείνετε ε, δημοκρατική δομή των εσωτερικών σας δομών. Άκουσα τι είπατε για τους ε, τραστείς και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά αυτό δεν αρκεί για να ανταποκριθεί στις αρχές της δημοκρατίας. Νομίζω ότι η απάντηση Βεβαίως και δεν είμαστε ταυτόσιμοι με μια κεντρική τράπεζα, αλλά θεωρώ ότι χρειαζόμαστε την ανεξαρτησία μας, διότι δημιουργούμε πρότυπα τα οποία έχουν μεγάλη επιρροή στις επιχειρήσεις και ε, στο παρελθόν σε πολλές χώρες ε, ε, ο καθορισμός των προτύπων ήταν εγγενής του ιδιωτικού κλάδου και εξακολουθεί να είναι σε κάποιες περιπτώσεις και ορισμένες φορές αυτοί που καθορίζουν πρότυπα έχουν και παράπλευρα καντεθήκοντας στον ιδιωτικό κλέδο. Για μας αυτό είναι αναπόφευκτο. Παραδείγματος χάρη, θέλουμε να δημιουργήσουμε τώρα ένα πρότυπο, μια προδιαγραφή και υπάρχει μεγάλη αντίθεση από τον ιδιωτικό κλάδο γιατί θέλουν αυτά τα πράγματα να μην περιλαμβάνονται στους ισολογισμούς των επιχειρήσεών τους. Για μας είναι πολύ σημαντικό όμω να τα καταφέρουμε αυτά και αν δεν υπάρχει ανεξαρτησία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πολύ πιο δύσκολο ε, αυτό. Επομένως, ναι, ε, είναι ιδιωτικό ο ρόλος μας, δεν είμαστε ρετοί, ε, δεν εκλεγόμαστε με δημοκρατικό τρόπο, δεν ξέρω εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να εκλέγει λογιστές, αλλά δεν εκλέγεται όλα τα μέλη των Ευρωπαϊκών ε, Δημοσίων Οργανισμών, ούτως ή άλλως. Ε, Πολλό δε μάλλον, εσείς δεν είστε λογιστές, είστε αυτοί οι οποίοι καθορίζετε τις πραδιογραφές, τα λογιστικά πρότυπα και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν είστε λογιστής είστε αυτοί που καθορίζετε τα πρότυπα για τα λογιστικά και είναι πολύ μεγάλη διαφορά και το επιχείρημά σας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τομείς της οικονομικής πολιτικής. Επομένως δεν υπάρχει κάποια αιτιολόγηση ε, για το γεγονός ότι δεν εκλέγεστε. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Ε, κοιτάξτε, εάν τα κράτη-μέλη του IASB, του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, που χρησιμοποιούν τώρα τα πρότυπά μας, θεωρούν στο μέλλον ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας οργανισμός που να καλύπτει από κάποια τέτοια σύμβαση, ε, το θα πρέπει να γίνει. Προς το παρόν δεν ε, γίνεται κάτι τέτοιο γιατί δεν χρησιμοποιούνται από όλου τα πρότυπά μας. Θα ήταν πολύ περίπλοκο ούτως ή άλλως να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, προς το παρόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος βαθμός ανεξαρτησίας προκειμένου να προστατευτούμε από τα εμπορικά συμφέροντα. Και αυτό κάνει ο οργανισμός μας. Σε ευχαριστούμε. Από εσάς υπάρχει κάποιος ομιλητής, όχι. Μπερνά Μονό, επόμενος αγορητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η διακυβέρνηση είναι στον πυρήνα των συζητήσεων μα για τα λογιστικά πρότυπα, Όμω πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ε, δεν παρεμβαίνει σε μεγάλο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ρυθμιστική διαδικασία θέσπιση δηλαδή νέων προτύπων. Από την άλλη πλευρά ε, υπάρχει και ο ρόλο των μεγάλων ελεγκτικών οργανισμών ε, στα πλαίσια τη ISP. Το είπε και ο κύριο Μέισταντε και όταν ανέλαβε ο, κύριο, ο Επίτροπος Μπαρνιέ μίλησε για την διακυβέρνηση της ISB και είπε, ISB συγγνώμη, και είπε ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Ε, το, μίλησε για την επιρροή του αγγλοσαξονικού μεντόλου και ανέφερε ότι πρόκειται για το όριο της, ε, των ε, διεθνών προτύπων διότι ακολουθείται μια λογική βράχη πρόθεσμη, κοντόφθαλμη ε, που στρέφεται προς τη λειτουργία των αγορών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς βλέπετε το μοντέλο της ISB ε, ε, και κυρίως ως προς την εκπροσώπηση των εθνικών μελών και κυρίως του ευρωπαϊκού τμήματος. Επίσης, μακροπρόθεσμα, πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πρότυπα για να τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη, πιστεύετε ότι εξυπηρετούν ουσιαστικά τις αγορές και οι επιχειρήσεις ε, τελικά αντί να υιοθετούν μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές τρέφονται προς ε, βραχυπρόθεσμες επενδυτικές πολιτικές με σκοπό το άμεσο όφελος. Για την πρώτη σας ερώτηση λοιπόν ποιες εξελίξεις σε σχέση με τη διακυβέρνηση θα ήθελα να ενθαρρύνω ήδη το προανέφερα ότι αυτή τη στιγμή περίπου δύο τρίτα των ε, εσόδων μας είναι από ε, δημόσιες ε, πηγές χρηματοδότησης και έχουμε ακόμα και κάποια έσοδα από ιδιωτικές πηγές. Η ιδέα και ιδανικό μας θα ήταν στο μέλλον να είναι μόνο από δημόσιες πηγές όλα μας τα έσοδα και υπό την επιτήρηση και εποπτεία των, του ε, χρηματοοικονομικού ε, οργάνου. Υπό την πτυχή της μακροπρόθεσμης πτυχής επενδύσεων, πρώτα απ' όλα, συχνά μας κατηγόρησαν κατά το παρελθόν ότι είμαστε φετιχιστές των αγορών και ότι όλα βασίζονται σε σχέση με αξίες και τιμές αγοράς. Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Έχουμε ένα μεικτό πρότυπο και οι λογιστικές μας πράξεις βασίζονται ιδιαίτερα για την μη χρηματοοικονομική πτυχή ε, σε πτυχές, σε ε, πρότυπα λογιστικά αξιόπιστα. Οι ε, λογιστικές αυτές προσεγγίσεις θα δημιουργούσαν μια τεχνητή ε, μεταβλητότητα, μεταβλητότητα που δεν θα ήταν ιδανικό ε, στοιχείο για την αγορά. Το καλύτερο για την παροχή διαφάνειας που θα εμπιστευόντουσαν αυτοί οι επενδυτές είναι αυτό το μεικτό σύστημα το οποίο παρακολουθεί τις πραγματικές εξελίξεις εκ του σύνεγγης και είναι η καλύτερη εγγύηση που μπορούμε να δώσουμε για τις μακροπρόθεσμες ε, επενδύσεις και επενδυτές διότι αυτό είναι κάτι το κεκτημένο και ε, ιδιαίτερα σημαντικό για τις ε, επιχειρήσεις. Θα προσθέσω κάτι για τη σύνθεση του Συμβουλίου και την ε, πολιτισμική επιρροή. Λοιπόν, για το σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουμε ένα Βραζιλιάνο, ένα Κορεάτη, έναν Κινέζο, έναν Νοτιοαφρικανό, πέντε Ευρωπαίους, τρεις Αμερικανούς, δύο Ασιάτες, δεν έχω την εντύπωση ότι είναι ε, υπερβολική πολιτισμική επιρροή του αγγλοσαξονικού τρόπου σκέψης στο Διοικητικό Συμβούλιο, μόνο και μόνο από τη σύνθεση. Ωραία. Να περάσουμε τώρα στο Catch the Eye. Σιλβί Γκουλάχ. Ευχαριστώ. Το ερώτημα του Σφεν Γκίκολ μου φαίνεται πολύ σημαντικό. Ε, δεν έχουμε τίποτα εναντίον σας. Ε, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Και το ίδιο ρώτησα στον ε, κύριο Καρονέ από την Επιτροπή της Βασιλείας της, του Διεθνούς Οργανισμού Συμψηφισμού. Έχουμε πρόβλημα διότι θεσπίζονται τα πρότυπα, αυτά τα πρότυπα που επηρεάζουν πολύ σημαντικά την οικονομία και θεσπίζονται εκτός κάθε δημοκρατικής διαδικασίας. Στα πλαίσια του G20 μιλάμε φυσικά για την διεθνή διεθνή συνεργασία ε, και έχουμε πλήρη επίγνωση ότι χρειαζόμαστε διεθνή συνεργασία. Ναι, όντω, όμω αυτό πρέπει να είναι ει βάρο του δημοκρατικού ελέγχου. Μπορούμε δηλαδή να συνεχίσουμε να δεχόμαστε να συμβαίνουν αυτά χωρί διάλογο. Ε, και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ή να εκμηδενήσω ε, αυτά που κάνετε, να παρακάμψω το έργο σας, ε, τι σκοπεύετε να κάνετε για να επαναφέρετε το θέμα της υιοθέτησης των νέων προτύπων στην καρδιά του δημοκρατικού διαλόγου, της δημοκρατικής διαδικασίας. Απάντηση. Όπως είπα και προηγούμενα, θα μπορούσα να το φανταστώ, αλλά μέχρι σήμερα δεν ήταν σημασίας σημασία σπουδαιότητα θέμα Ίσως στο μέλλον οι αδερφές οργανώσεις μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν αυτές, αυτά τα πρότυπα για την αλλαγή διακυβέρνησης αν θα το επιθυμούσαν ή αν θα ήθελαν να είναι μια, ε, ένα σύνολο με βάση μια συνθήκη. Η συμφωνία είναι περίπλοκο εγχείρημα αυτό. Αυτό το οποίο άλλαξε μέχρι σήμερα στο πρόσφατο παρελθόν είναι τούτο. Το ότι κατά το παρελθόν σε σχέση με, μια, με την απουσία του επι, ε, εποπτικού οργάνου. Τώρα έχουμε ε, ε, την εποπτεία, την επιτήρηση και αυτό τουλάχιστον έχει διασφαλίσει ένα, μια δημόσια παράμετρο σε σχέση με το όργανό μας και αυτό είναι σημαντικό. Λυπούμε πολύ το πρόβλημα δεν είναι να υπάρχει μια συνθήκη ή να υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο, αλλά η δημοκρατία και η δημόσια συζήτηση και λογοδότηση. Τι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε εμείς ε, τα αιτήματά μας, ε, θα μπορούσατε να εισακούσετε εσείς τα αιτήματα αυτά. Το δικό σας όργανο δεν εργάζεται δημοκρατικά. Να υποβάλλετε προτάσεις, να ενεργοποιηθείτε περισσότερο για να βελτιωθούν τα πράγματα. Πολλά πράγματα είναι περίπλοκα στην ε, καθημερινή ζωή, αλλά τα θέματα δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Δεν γνωρίζω τι σημαίνει εδώ η όρος δημοκρατία, αλλά πραγματικά προσπαθούμε να είμαστε όσο ανοιχτοί και όσο διαφανείς γίνεται σε σχέση και με τα πρότυπά μας. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Έχουμε πολλές συμβουλευτικές επιτροπές. Υπάρχει μεγάλη συνεισφορά από πλευρά ε, της Ευρώπης. Ε, είμαστε λοιπόν μια πολύ ενεργό σε αυτά τα πλαίσια ε, οργάνωση. Μπερές, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στη Monitoring Group, αλλά επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω από που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία. Προήλθε σε συνέχεια μια έκθεση του κυρίου Ράτβαν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, μια ανησυχία η οποία κορυφώθηκε και από πλευράς του αρμοδίου ε, επιτρόπου τότε, ήταν ο Τσάρλι Γκρίβι και υπήρχε και ο κύριος Τουίτη, ο οποίος ανησυχούσε επίσης και αμφισβητούσε τον τρόπο διακυβέρνησής σας. Και τότε επιγόντως κινητοποίησαμε και τους Αμερικανούς και τους Ιαπωνέζους. Ε, ε, οι Αμερικανοί δεν είχαν ε, και καμία δουλειά, δεν, ασχολ... δεν εφαρμόζουν τα IFRS, ούτε τότε ήθελαν να τα εφαρμόσουν και συστάθηκε αυτή η monitoring group. Και μετά από κάποια χρόνια βλέπετε ότι ο βαθμός της δυσαρέσκειας εξακολουθεί να είναι περίπου ίδιος. Δεν βελτιώθηκε και πολύ και ε, ε, εγώ λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η ομάδα, η monitoring group και υπάρχει για δύο λόγους κατά την άποψή μας. Από δημοκρατική σκοπιά καταρχάς, ότι δεν, διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι ένας λογιστικός κανόνας είναι απλώς ε, ένα τεχνικό ζήτημα. Πες μου τι γράφεις και θα σου πω τι εννοεί. Ε, και το λογιστικό πρότυπο ε, είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια των στοιχείων ούτε των προτύπων, διότι εάν υπήρχε η απόλυτη αλήθεια δεν θα υπήρχε τόσο ανάγκη να σπαταλάτε τόσο χρόνο να τους ετοιμάσετε. Θα πρέπει να επιλέξετε ποιο μοντέλο ευνοείται και κατά την κατάρτιση αυτών των προτύπων ε, Υπάρχει και το θέμα της σχέσης με τις δημόσιες αρχές, όχι πέρα, πέραν της χρηματοδότησης, πρέπει φαίνεται ότι αυτό που θέλουμε συλλογικά είναι ε, αυτό το οποίο υπερτερεί σε σχέση με αυτό το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει. Και το θέμα είναι τι γίνεται με τις ε, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Εμένα πολύ συχνά οι επενδυτές οι οποίοι κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις μου λένε ότι δεν μας επιτρέπεται να έχουμε καλές συνθήκες ε, επένδυσης μακροπρόθεσμες. Και ξέρω ότι δεν είστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να βελτιώσετε την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση, αυτό είναι αποδεκτό βεβαίως, αλλά θεωρείτε ότι υπάρχει τρόπος να εισακουστεί η φωνή των Ευρωπαίων. Διότι ορισμένες φορές φαίνεται ότι κάποια πράγματα προκύπτουν περισσότερο λόγω της δικής σας της ανησυχίας και όχι λόγω της ανησυχίας των Ευρωπαίων. Και ένα τελευταίο, αφού έχω το λόγο, πέραν του δημοκρατικού ζητήματος, ε, γιατί ε, ξεκινάτε να καθορίσετε το τάδι το δίνα πρότυπο. Το σύστημα της νομοθεσίας σε χρηματοοικονομικά ζητήματα, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να είναι ευθύνη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εσείς είστε ένας οργανισμός απόλυτα ανεξάρτητος, με ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο έχετε ρυθμίσει εσείς, έχετε φεύρει μόνοι σας ουσιαστικά για να μην υπάρχει ανάγκη να ε, συμμετέχετε σε κάποιο σύνολο. Και θεωρώ, εξακολουθώ να θεωρώ ότι αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα τα οποία δεν έχει διασκεδάσει σε καμία περίπτωση η σημερινή σας παρέμβαση εδώ. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να επαναλάβω για άλλη μια φορά η Ευρώπη δεν αγκατέλειψε, δεν απεμπόλησε τα κυριαρχικά της δικαιώματα επ' αυτού. Στο, στο τέλος τέλος πρέπει να βελτιωθούν σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο τα πρότυπά μας και οι προδιαγραφές μας. Αν είσαστε δυσαρεστημένοι λοιπόν σε σοβαρό βαθμό μπορεί να αρνηθείτε, μπορείτε να αρνηθείτε αυτά. Είναι ένα είδος πυρηνικού όπλου αυτό, αλλά μπορώ να σας δώσω, δίνει στην Ευρώπη μεγάλη μόχλευση και σε σχέση με τους ε, ε ως εμπλεκόμενους στην παγκόσμια σκηνή Καμιά φορά αισθάνονται ότι έχουν υπερβολική μόχλευση και επιρροή οι Ευρωπαίοι λόγω αυτής ακριβώς της δυνατότητας που ε, ενυπάρχει στην Ευρώπη. Και δεν απηχούνται οι δικές μας, τα δικά μας ε, μελήματα σε σχέση με την ΙΦΡΕΚ. Έχουμε έντονο διάλογο και πολλές φορές διαφωνούμε σε σχέση με τις απόψεις τους. Ε, το πλήρες ε, πρότυπο των ε, λογιστικών προτύπων δεν είναι απόλυτη εγγύηση επιτυχίας και επιτρέψτε μου να επαναλάβω αυτό το οποίο ανέφερα στις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις πολύ μεγάλος βαθμός ε, από τις δημόσιες δραστηριότητες σε σχέση με τα πρότυπα αυτά έχουν κενά και ελλείψεις και δεν υπάρχει πλήρης εικόνα. Και αν ήταν όλα αυτά ανάγλυφα εξόφθαλμα όπως σε σχέση με τις ε, προδιαγραφές που ισχύουν τώρα σε σχέση με μας, θα ήταν πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα τα οποία θα αποκαλύπτονται. Δεν είναι λοιπόν εγγύηση αυτό αυτού. Ευχαριστώ. 10 seconds. δευτερόλεπτα εσείς. Μα δεν ρώτησα αυτό. Αυτό που είπα να διασφαλίσουμε ότι με τα δικά σας πρότυπα να υπάρχει η χρηματοοικονομική σταθερότητα που θα λαμβάνετε υπόψη. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει εντονότερη διασύνδεση σε σχέση με τα τεκτενόμενα από πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όπως σας είπα, είμαι μέλος ε, του ε, Συμβουλίου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας και το θεωρώ ως δική μας ευθύνη επίσης να συνεισφέρουμε υπέρ της χρηματοοικονομικής ε, σταθερότητας και πιστεύουμε ότι η διαφάνεια είναι τεράστια συνεισφορά για τη σταθερότητα. Πριν από την χρηματοοικονομική κρίση εξετάζοντας τους ισολογισμούς των τραπεζών θα μπορούσε κανείς να δει ότι δεν είχαν κεφάλαια οι τράπεζες αυτές. Ήταν ε, λοιπόν εξόφθαλμο και μπορούσε κανείς να το δει αυτό, αλλά επέλεξαν κάποιοι να μην το δουν και να μην το εντοπίσουν. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που έχουμε λοιπόν να διαδραματίσουμε, συμφωνώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη και ζωντανή αυτή η συζήτηση και αν μου επιτρέπουν οι συνάδελφοι θα έλεγα ως συμπέρασμα ότι είναι σαφές ότι αυτή η κοινοβουλευτική μας επιτροπή έχει κάθε λόγο κιόλα. να πει ότι πιθανότατα υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις κιόλα και για την δημοκρατική λογοδοσία στο έργο ακριβώς που επιτελείτε εσείς. Όμως να λάβουμε επίσης υπόψη και τούτο, το ότι έχουμε ισχυρά μέσα και εργαλεία που θα έπρεπε στο πλαίσιο της έκθεσης Σιλβί Γκουλάρ να δούμε πώς μπορούμε πιο αποτελεσματικά να τα χρησιμοποιήσουμε. Εκλέγουμε την Επιτροπή και τα μέλη του Συμβουλίου. Τώρα θα εκλέξουμε το νέο πρόεδρο ΕΦΡΑ και θα δημιουργηθεί μια νέα σχέση λογοδότησης υπεύθυνων σχέσεων με την ΕΦΡΑΚ. Και έτσι λοιπόν σε σχέση με τη λογοδοσία θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι απαιτήσει μας. Έχουμε επίσης και τον προϋπολογισμό και έχουμε επίσης τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και από πλευράς επιτροπολογίας και καθώς βλέπουμε με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις πολλά μπορούν να επιτευχθούν για να υπάρξει μια πιο ισχυρή σχέση στην ε, προληπτική φάση των πραγμάτων. Είναι σαφές ότι το πυρηνικό όπλο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς αν το αποφασίσει, αλλά δεν είναι καθημερινής χρήσης. Με την έφραχη λοιπόν εμείς, εμείς ε, Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να πούμε εμεί οι ίδιοι στον εαυτό μα, όχι σε εσά. Να το λέμε σε εμά. Μπορούμε καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα και εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα για να έχουμε μια πιο ζωντανή και ισχυρή σχέση μαζί σα και με την ΕΦΡΑΚ. Ήταν χρήσιμη λοιπόν αυτή η συζήτηση σίγουρα και πιθανότητα μέσα στο πλαίσιο αυτό τη έκθεσή μα, έκθεση Γκουλάρ, θα μπορέσουμε πιθανότατα να επισέλθουμε σε μεγαλύτερο βάθος σε αυτά τα θέματα και σε διάλογο και επαφή μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Και περνάμε στη συνέχεια στο επόμενο θέμα, στην ημερήσια διάταξη. Ο κανονισμός για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς. Έκθεση Νίνα Τζιλ. Έχουμε ε, σχέδιο έκθεσης όπου γίνεται μια νέα πρόταση σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, φαντάζομαι θα γίνει ζωντανή συζήτηση ζωηρή συζήτηση και για αυτό το ζήτημα. Νίνα, παρακαλώ, σας ακούμε. Να ξεκινήσω λοιπόν πρόεδρε υπενθυμίζοντας τους συναδέλφους για τη χρονική παράμετρο. Από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων τον Οκτώβριο 13 Οκτωβρίου είχαμε μία στρογγυλή τράπεζα, μία βίντεο διάσκεψη και πάμπολες συναντήσεις ε, με το ρυθμιστικό τομέα και μια ευκαιρία επίσης πάλι να συναντήσουμε και τους σκιώδεις εισηγητές, να συναντηθούμε. Κατέθεσα σε 11 Νοεμβρίου το σχέδιο εκθεσής μου. Θα δείτε από αυτό ότι οι κύριες ανησυχίες και μελήματά μου ήταν πώς να αντιμετωπιστούν οι συστημικοί κίνδυνοι σε σχέση με αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια αγορα, χρήματα δεν θέλω τώρα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία να επαναλάβω τα πάντα και να επισέλθω σε λεπτομέρειες τι είναι αυτές ε, οι αγορές ε, ε, αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς. Θέλω όμως από την άλλη πλευρά να υπενθυμίσω σε όλους γιατί βρισκόμαστε εδώ και γιατί έχουμε αυτή την έκθεση ενώπιόν μας. Διότι δυστυχώς πολύ σημαντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει κατά τη διάρκεια της κρίσης και από την πτώση των Lehman Brothers πάρα πολλά συνέβησαν στο χρηματοοικονομικό τομέα. Καθώς επίσης ε, και όσον αφορά τα ε, ταμεία αυτά. Επίσης ε, για τις κατευθυντήριες γραμμές 2010 για ορισμούς και τύπου πολιτικών που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε το Σεπτέμβριο 2013 την πρότασή της ως επόμενο βήμα. Εμείς ε, εφέτος το καλοκαίρι υιοθετήσαμε μια ευρύτερη μεταρρύθμιση του κανονισμού. Ο στόχος μου ήταν ε, να αντιμετωπιστούν οι συστημικοί κίνδυνοι όπως προανέφερα σε σχέση με αυτές τις ε, χρηματοοικονομικές αγορές και να δούμε κατά κάποιο τρόπο πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πρώτον για τις απαιτήσεις ρευστότητας που είναι στο άρθρο 21 και στο άρθρο 22 που προτείνουν να αυξηθούν από 10% ρήμανση σε 20% ρήμανση αυτά τα αποθέματα και τα εβδομαδιαία από 15% σε 30%. Όσο μεγαλύτερη ρευστότητα αυτών των ταμείων, τόσο πιο εύκολο θα είναι να πωλήσουν αυτά τα το δυναμικό που διαθέτουν. Και έτσι λοιπόν θα, είναι πιο, ε, θα υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια. Και επίσης στο άρθρο 15 για την πολυμορφοποίηση που προτείνουν να ενισχυθούν αυτές οι διατάξεις. Διότι πολλά προβλήματα απορρέουν όταν οι αγορές εξαρτώνται υπερβολικά από μία παράμετρο. Γι' αυτό προτείνω να μειωθούν αυτές οι απαιτήσει από 10% σε 5%. Και όσον αφορά την ε, ε, ανταπόκριση που μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την ε, ρευστότητα. Και σε σχέση με τα όσα έχουν προβλεφθεί στο άρθρο 35, διότι είναι προφανές ότι στο παρελθόν κάποια ταμεία μπορούσαν να παραμείνουν ενεργά μόνο λόγω γενναιόδορης υποστήριξης από τις τράπεζες που τα υποστήριζαν δισεκατομμύρια που δόθηκαν σε αυτά τα ταμεία από το 2007 στο 2011. Δεν είναι ιδανική καθόλου αυτή η κατάσταση δεδομένου του μολυσματικού χαρακτήρα των συστημικών κινδύνων και υπάρχει κίνδυνος να διαδοθεί αυτό, αυτή η μόλυνση ε, στον τραπεζικό τομέα. Και εδώ λοιπόν σε σχέση με τις ε, διατάξεις που θα πρέπει να ε, λειτουργούν, αν δεν λειτουργήσουν θα υπήρχε μείζον πρόβλημα και θα είχε αυτό τεράστια επίπτωση όσον αφορά τους ε, ισολογισμούς αυτών των τραπεζών. Η μόνη λοιπόν εξαίρεση που θα δεχόμουν θα ήταν να χρηματοδοτείται το κεφάλαιο κινδύνου. Ωστόσο, οι ρυθμιστές θα πρέπει να εγκρίνουν τέτοιου είδους υποστήριξη από πλευρά Τέταρτον, ζητώ να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια αυτό για μένα είναι ένας τρόπος να περιοριστούν οι κίνδυνοι και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι περιοδικές μόνο οι αναφορές και οι εκθέσεις όσον αφορά την υλοποίηση των απαιτήσεων, αλλά θα έχουμε ένα τριμηνιαίο διάστημα τέτοιες εκθέσεις και αξιολογήσεις και τα ταμεία αυτά θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι πιο εξειδικευμένα θα αναφέρουν όσον αφορά τη ρευστότητά τους, την ανταγωνιστικότητα που διασφαλίζουν και τον ανταγωνισμό όσον αφορά τις ε, επενδυτικές δραστηριότητες. Και για τις επιλέξιμες δράσεις ε, περιόρισα το φάσμα και σε σχέση με τα παράγωγα διότι θεωρώ ότι πρέπει να είναι πιο συνετό το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργούμε να μειώνονται οι κίνδυνοι από πλευράς των παραγόγων και έτσι να βελτιώσουμε την διαχείριση αντιμετώπισης κινδύνων. Τρίτον, προσπάθησα να ενισχύσω την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι πεισμένη ότι θα έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα μέσα, αυτά τα ταμεία θα είναι ένα μέσο της πραγματικής οικονομίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μειωθεί το εύρο συζήτηση για τα ταμεία αυτά μόνο σε κάποιες πτυχές. Ακούσαμε όλοι τον πρόεδρο Γιούγκερ να λέει ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα στις επενδύσεις ε, για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε ότι δεν έχουμε μόνο το θέμα της ε, βραχυπρόθεσμης επένδυσης αλλά μακροπρόθεσμα πρέπει να μπορέσουμε και να δράσουμε και για το συστημικό κίνδυνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί να δούμε αν θα είναι με, την, ε, το πλαίσιο της ε, SNAV, SNAV ή VNAV. Δύο διαφορετικά μέσα προτάθηκαν ε, σε σχέση δηλαδή με τις σταθερές ΚΑΕ και τις μεταβλητές ΚΑΕ. Και εδώ έχω και τις απόψεις μου, έχω και κάποιες επιφυλάξεις, παρότι κατανοώ βέβαια πώς καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα οι συνάδελφοι και σε κάποιες προτάσεις. Σε σχέση με τη ρευστότητα, είναι μια πρόταση που υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις. Δεν είμαι βεβαία ότι αντιμετωπίζονται οι συστημικοί κίνδυνοι όπως εγώ θα ήθελα να αντιμετωπιστούν. Έχω επίσης επιφυλάξεις όσον αφορά το κεφαλαιακό ε, μαξιλάρι ή απόσβεση κραδασμών, buffer, ε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι, έχω πιστεί ακόμα ότι αυτή η διατύπωση είναι η σωστή απάντηση για την μετατροπή δηλαδή του συνάβα το ΒΙΝΑΒ ε, για την ε, διασφάλιση των παραμέτρων της αγοράς όταν κάνουμε λόγο για ε, δισεκατομμύρια. Επίσης θα μπορούσαν πολλές φορές να οδηγηθούν κονδύλια σε ιδιωτικές επενδύσεις ιδιωτελώς που θα βρισκόντουσαν εκτός ελέγχου. Προσπάθησα μια εναλλακτική λύση να εκπονήσω συλλέγοντας στοιχεία από διαφορετικές προσεγγίσεις. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ μείζον πρόβλημα σε σχέση με το βαθμό συνεκτικότητας και συμβατότητας μεταξύ διαφορετικών ε, δυνατοτήτων ρυθμίσεων. Με τρεις τύπους ε, δυνατοτήτων ε, παρέμβασης στις αγορές. Πρώτον, τον τομέα Βίναβ. Και δεύτερον, το δημόσιο, τον συσχετισμό σε σχέση με το δημόσιο χρέος, χρέος του Βίναβ. Και αν υπάρχουν προβλήματα θα υπάρχει εναλλακτική λύση για να ενταχθεί κάποιο στο πλαίσιο ΒΙΝΑΒ ή να αναζητηθεί μια εναλλακτική λύση σε σχέση με επενδυτικά προϊόντα. Επιτρέψτε μου να επισέλθω σε σχέση με τη ΣΥΝΑΒ σε κάποιες παραμέτρους μπορεί να παραμείνουν σε αυτό το πλαίσιο εφόσον κατά το 2020 το 80% των, ε, αποθεμα... Ε, ε, του δυναμικού τους θα βρίσκονται σε συσχετισμό με τις χρεωστικές πράξεις. Αν δεν επενδύονται στο δημόσιο χρέος τότε θα υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι 3% που μέχρι το 2020 θα μπορεί να αναπτυχθεί και που μπορεί να συνυπολογιστεί σε σχέση με τους κινδύνους και να μπορέσει έτσι να αντιστοιχεί στην δυνατότητα αυτή. Ε, έτσι αναφερόμαστε λοιπόν σε αυτό το μαξιλάρι στην αναλογία ε, capital buffer από θεματικό ασφάλειας και να δούμε κατά πόσον θα πρέπει να αναπτυχθούν ε, δυνατότητες ώστε να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για τα κεφάλαια ασφαλείας. Πιστεύω ότι Αυτά τα ταμεία ΒΙΝΑΦ μπορούν να συνεισφέρουν ε, ώστε να συνεισφέρουν με για τη χρηματοδότηση της πραγματικής ε, ευρωπαϊκής οικονομίας. Να αντιμετωπιστούν βραχυπρόθεσμα οι προκλήσεις για τις επενδύσεις. Δέχομαι ότι αυτή η ιδέα δεν είναι ε, ελευθέρα κινδύνου, δεν απουσιάζουν οι κίνδυνοι από αυτή την πρόταση. Απόλυτα πιστεύω ότι πρέπει να δοθούν ευκαιρίες ώστε να προσαρμοστούν τα κεφάλαια αυτά ε, στην πραγματικότητα και πρέπει με πολύ, ε, σταδιακό, με πολύ βήμα προς βήμα σταδι, σταδιακή εξέλιξη ε, να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε αυτή την προσαρμογή. Μία πρώτη αξιολόγηση μετά από τρία χρόνια θα μπορούσε να γίνει και να δούμε πώς είναι δυνατόν να αντιστοιχείτε στο χρέος. Γι' αυτό θέτουμε ένα όριο αναεκδότη. Δεχόμαστε ότι η αγορά είναι πολύ μικρή. Αυτή τη στιγμή 60 με 65 δις ευρώ συνολικά. Και συμφωνώ από την άλλη πλευρά ότι αυτή τη στιγμή μια και έχουμε ένα 12% περίπου των δημόσιων χρεογράφων που είναι ε, μικτού χαρακτήρα ε, ε και ΙΠΑ. Αν δείτε όμως τη σελίδα 67 της μελέτης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προαναγγέλλεται ότι μπορεί ταχύτερα να επιτευχθεί ανάπτυξη και να υπάρξει μια εναλλακτική δυνατότητα προσαρμογής. Η Βίναβ ε, έχει, βρίσκεται υπό συζήτηση και ήρθαν σε επαφή μαζί μου και μου είπαν ότι μέχρι, μέχρι το ένα συγκεκριμένο ποσοστό επενδύσεων θα μπορούσε να διασφαλιστεί. Δεν βλέπω καν να υπάρχει κάτι το αρνητικό στο να προσπαθήσουμε να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι μέχρι το 2020 για το ποσοστό αυτό αναφέρθηκαν όλοι οι λόγοι γιατί οι εναλλακτικές δυνατότητες ε, μετατροπής στο ΒΙΝΑΦ ε, δεν θα ήταν αποδεκτές. Νομίζω τους προσφέρεται μια δυνατότητα για μια στρατηγική ανάπτυξης ε, και απασχόλησης. Και όπως είπα υπάρχουν πολλά ωφέλη από αυτό το εγχείρημα. Ένα από αυτά θα ήταν το ότι το κυβερνητικό χρέος ε, θα είχε υψηλή ρευστότητα χαρακτήρα και θα μπορούσε να επωφεληθεί από τις βραχυπρόθεσμες δράσεις ε, και θα μπορούσε να διασφαλίσει υψηλού επίπεδου πιστώσεις. Ε. Ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι γνωρίζω ότι οι επιχειρήσεις θέλουν να έχουν μια εναλλακτική δυνατότητα επενδύσεων στο χρέος των ήπα Δεν ε, συμπεριέλαβα αυτή την εναλλακτική δυνατότητα και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στην οικονομία της ΕΕ και όχι στην οικονομία των ΗΠΑ. Αν ε, θα ήταν αυτό κάτι στην αναθεώρηση και επανεξέταση που θα μπορούσε να τύχει προσοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν θετικό. Στρεφόμενοι τώρα στο συστημικό κίνδυνο, συστημικούς κινδύνους στη ΣΥΝΑΒ, αναφερόμενοι στην κρίση 2008-2011 καταδείχθηκε ότι οι κυβερνητικές αυτές δυνατότητες όταν ένα ταμείο αντιμετώπιζε δυσκολίες θα, μπορούσε να θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα ασφαλή λιμένα διαθέτοντας έτσι κονδύλια από τη μία πηγή στην άλλη θα έπρεπε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ασφαλούς λιμένα. Ενώ γνωρίζω απόλυτα και αξιολογώ το ότι δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση και δεν αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση όπως είπα, δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε μια τέτοια προσέγγιση, θα έπρεπε να εξετάσουμε δυνατότητες και ίσως να ενθαρρύνουμε ένα τέτοιο πρότυπο προσέγγισης και να δούμε ότι το κεφαλαιακό, οι κεφαλαιακές δυνατότητες δυνατότητες ε, ασφάλειας ε, δεν είναι πάντα δεδομένες, ε, το αποθεματικό ασφάλειας δηλαδή. Και να δούμε τους κινδύνους που υφίστανται και να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στη συνολική αξία επενδύσεων. Όμως ε, όταν έχουμε περίοδο χαμηλών επιτοκίων όπως ε, σήμερα σε αυτή τη συγκυρία πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί. Αυτά τα κονδύλια χρειάζονται, αυτά τα χρήματα ε, πιο μακροπρόθεσμα. Βρίσκον, στρεφόμενοι τώρα στην λιανική αγορά κατά τη διάρκεια της κρίσης είδαμε ότι μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές είχαν δραστηριοποιηθεί και όχι μικρότερων διαστάσεων, μικρότερης εμβέλειας επενδυτών που ήταν τα θύματα περισσότερο και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από αυτά τα θεσμικά ε, όργανα δεν επιτρέπεται σε κειμενόμενες, ε, ε, ισχυρά κειμενόμενες αξίες να επενδύουν, θα έπρεπε να μπορέσουν να εξαιρεθούν και να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο. Αν δει κανείς λοιπόν το, τα 82 δις, για παράδειγμα, σε σχέση με την Λιανική αγορά και τις επενδύσεις. Συμφωνώ απόλυτα και το ε, εκτιμώ ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ορισμών. Όμως δεν είναι στόχος μου να ανοίξω πόρτα και παράθυρο ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτός ε, δυνατότητα εξαίρεσης ώστε όλοι να θεωρούνται μετά ε, εμπλεκόμενοι στο πλαίσιο λιανικής. Γι' αυτό εξέτασα το παράτημα 2 του MIFID όσον αφορά ειδικού επενδυτές και αυτό είναι εκείνο το οποίο θα θέλαμε να ενταχθεί ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια από πλευράς ορισμών ενώ τα περισσότερα τα οποία προτείνω βασίζονται σε γεγονότα και αριθμητικά στοιχεία τα οποία ήταν διαθέσιμα και δημοσιεύθηκαν ε, τον ε, προηγούμενο Σεπτέμβριο ε, με την αξιολόγηση και συλλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συνοψίσω θέλω να πω ότι στόχος μου είναι να υπάρξει ισχυρή πολιτική συμφωνία τους επόμενους μήνες ώστε να υπάρξει μια ισόρροπη σχέση προστασία των κονδυλίων των φορολογουμένων, αντιμετώπιση των κινδύνων αλλά δημιουργώντας και δυνατότητες επενδύσεων για τις, τις οικονομίες μας, την οικονομία μας από την άλλη πλευρά. Είναι ένα σχέδιο λοιπόν έκθεσης στο οποίο υπάρχουν σαφώς τροποποιήσεις, αλλαγές, προσαρμογές που πρέπει να συζητήσουμε και να εξετάσουμε και υπάρχει και μια συνάντηση που έχουμε συμφωνήσει με τους κοιόδης εισηγητές όπου ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να τα πετύχουμε, να γίνουν αυτές οι αλλαγές και προσαρμογές. Τούτων λεχθέντων είχαμε μια αντιπαράθεση κατά την τελευταία κοινοβουλευτική θητεία των δύο πλευρών ή των δύο θα έλεγε κανείς απόψεων ε, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε με αυτό το κανονισμό, με αυτή τη ρύθμιση, διότι αν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, αν δεν μπορέσει να εξευρεθεί η μέση οδός, το πρόβλημα το οποίο θα υφίσταται θα είναι ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές και προσαρμογές και δεν θα υπάρχουν καθόλου κονδύλια για αυτές τις ε, ρυθμιστικές δράσεις. Πρέπει να το λάβουμε λοιπόν σοβαρά υπόψη αυτό. Δεν μπορούμε να μείνουμε μετακίνητοι. Υπάρχει πολύ υψηλό επίπεδο συστημικών κινδύνων που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου. Και αυτό μια και βρίσκεται ακόμα στο σχέδιο ε, σύνταξης, στο σχέδιο έκθεσης, είχαμε πολύ καλή σχέση και όλοι οι σκιώδεις εισηγητές ενεργά συμμετείχαν. Θέλω να τους ευχαριστήσω και να αναγνωρίσω αυτό και λέγοντας ότι καθώς κινούμαστε προς το μέλλον είναι σημαντικό να μην θεωρούμε ότι είμαστε διχασμένοι. Όχι, είμαστε το Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει να δούμε ενωμένοι αυτό τον κανονισμό ως ανεξάρτητο κοινοβούλιο και να μην ε, υπαναχωρήσουμε και επαναλάβουμε την ίδια αντιπαράθεση με την ίδια συζήτηση όπως κατά το παρελθόν. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου που έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της ώστε να σημειωθεί πρόοδος. Ευχαριστώ. Thank you. Now Θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές και θα ήθελα να πω και στους αδέλφους που θέλουν να μιλήσουν να σκόσουν το χέρι τους για να μπορέσουμε να τους περιλάβουμε και στον κατάλογο των υπολείπων αγορητών. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν στους κοιόδης εισηγητές να μιλήσουν από δύο έως τρία λεπτά. Καταρχάς στους κοιόδης εισηγητής του ΕΛΚ, ο Μπράιαν Hayes. Μπορεί να μιλήσω λίγο παραπάνω από δύο λεπτά, ε, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, διότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, ζήτημα, πολύ σημαντική έκθεση. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Ε, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, μια ε, συζήτηση τρογγυλής τραπέζης με το SEC και ε, πιστεύω και συμφωνώ μαζί της ότι θα ήταν χρήσιμο να καταλήξουμε σε πολιτική ε, συμφωνία αλλά δεν θα ήταν έντιμο να πούμε ότι καταλήξαμε ήδη. Και παρά το γεγονός ότι πλέον έχει συμπεριλάβει τρεις νέες προτάσεις στο μείγμα, που δεν ήταν στην αρχική πρόταση τις οποίες βέβαια θα πρέπει να εξετάσουμε πιο διεξοδικά θα πρέπει να τονίσω κύριε Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να ε, εξετάσουμε το θέμα αυτό αναλογικά και να το δούμε. Έχει δίκιο η συγγήτρια όταν λέει ότι έχει δύο χρόνια που το εξετάζουμε το ζήτημα, 1,5 χρόνο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής χρειάστηκαν έξι χρόνια περίπου. Ε, με ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο 700 σελίδων και πάρα πολλές αξιολογήσεις αντικτύπου ε, πριν καταλήξουν σε αποτελέσματα τον Ιούλιο φέτος. Και η ουσία αυτών των προτάσεων θα καλύψουν ε, αλλαγές μόνο 10% στις ε, ε, αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η βασική ένσταση που έχουμε με τις προτάσεις αυτές είναι ότι έχει πάρει ουσιαστικά αυτό το μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτειών και προσπαθεί να το επιβάλλει στο μοντέλο που έχουμε εμείς εδώ. Ε, και πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα ε, το μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτειών και το δικό μας. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι πρέπει να είμαστε αναλογικοί και να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα. Η βασική παρατήρηση νομίζω ότι έγινε στραγγυλή τράπεζα από την Ελίζα Φερέιρα όταν αναφέρθηκε στο συστημικό κίνδυνο. Και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και λίγο και το ιστορικό σωστά εδώ κύριε Πρόεδρε, διότι αυτό που πρέπει να επιλύσουμε όλοι είναι το, ο συστημικός κίνδυνος. Διότι κανένα ευρωπαϊκό αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματοβόρας δεν είχε ε, θέμα... Ε, ε αξία του αποθεματικού τη. Αν κάποιο έχει δολάρια, παίρνει δολάρια. Αν έχει ευρώ, ευρώ. Δεν είναι η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι κονδύλια τα οποία χρησιμοποιούνται από μεγάλε επιχειρήσει. Και αυτό το οποίο συνέβη στις Ηνωμένε Πολιτείες, όπως είπε η Κινίνα, συνεπία των, των όσων συνέβησαν με τη Lehman Brothers, ε, ήταν στο παράδειγμα του δολαρίου με δολάριο. Δεν είχε 50 ή 60% επιστροφή, δεν είχε 50 cent ή 60 cent ε, στο δολάριο, ήταν 99 cent στο δολάριο. Και δεν ήταν κανείς υπόλογος για το έλλειμμα. Ουσιαστικά έχουμε ένα παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προτείνουμε μία ριζοσπαστική αλλαγή σε αυτό που προτείνει η Νίνα. Ε, το να προτείνουμε ΣΥΝΑΒ και VNAV στην Ευρώπη, ε, όταν έχουμε ένα 3 ε, ευρώ επενδύσεων σε ένα πολύ μεγάλο τραστ μεγάλων επιχειρήσεων και πολύ μικρό ποσοστό ε, λιανικών ε, κεφαλαίων. Και γι' αυτό ακριβώς και η αναδρομική λύση που θέλουμε να εφαρμόσουμε πρέπει να είναι ανάλογη αυτό που κάνουμε. Και αυτό που εννοώ είναι, αν δείτε και την τροπολογία 22 που έχει προτείνει η Νίνα στο ε, άρθρο 1, στην ουσία θα καταστρέψει το 80% του κλάδου των ΣΥΝΑΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ολοκληρώσετε, λέει ο Πρόεδρος. Έχω πάρα πολλά να πω από αυτού. Ε, ξέρω, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε από αυτού, αλλά έκανα πολύ σκληρή δουλειά. Σας παρακαλώ δύο λεπτά ακόμα την ανοχή σας. Ναι, αλλά δύο λεπτά μας σας δώσω, έχουν δικαίωμα να μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Η βασική μου παρατήρηση είναι εξή. Τζογάρουμε με αυτή την πρόταση ψάχνουμε να βρούμε, ε, όπως είπε και ο κύριος Γιούνκερ, ο πρόεδρος Γιούνκερ, ε, μια λύση σε ε, κάτι το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί. Και αν έχουμε μια λύση που δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα, για μένα είναι λανθασμένη λύση. Αυτό, ε, αυτή είναι η απόψή μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καμάρας, χειόδης εισηγητής ECR. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την Νίνα Γκίρ για τις ε, ενδελεχείς σκέψεις και εξέταση που ε, υπέβαλε αυτό το θέμα. Πραγματικά είναι σημαντικό αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ επίσης που προσπαθήσατε να παρουσιάσετε, να δημιουργήσετε νέες ιδέες. Είναι σημαντικό να γίνεται κάτι τέτοιο. Επίσης και για τις προτινόμενες λύσεις που υποβάλλετε. Όπως είπε ο Μπράιν πιο πριν, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αν αναζητήσει κανείς λύσεις αλλού, Πρέπει επίσης να δούμε αν είναι έφθετες ή όχι για τις ανάγκες μας και τι είναι διαφορετικό ή όχι, αν έχουμε τις ίδιες αγορές και παρόμοια στοιχεία, αν έχουμε το ίδιο δημόσιο χρέος με τα ίδια χαρακτηριστικά και πού θα καταλήξει αυτό το εγχείρημα και για ποιο χρέος κάνουμε λόγο και ποια μέτρα τα οποία θα αναλάβουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να είναι υψηλή ποιότητα ε, τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε. Αλλά επίσης και σε σχέση με ε, την λιανική αγορά, σε σχέση με τις ε, άλλες δραστηριότητες. Και επίση, πώ προέρχονται όλα αυτά. Αυτά ξεκίνησαν από το, μια εταιρεία για παράδειγμα που έχει υπόψη της να αγοράσει να, ε, μια, μια, μια παραγγελία ενός δισεκατομμυρίου και για το πώς θα μπορέσει να πληρωθεί αυτό παρά μόνο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Προστρέχει σε μια τράπεζα. Η δυνατότητα είναι να δοθεί ένα δισεκατομμύριο ε, ε, δολάρια και η συνεννόηση που θα γίνει θα είναι να ε, δοθούν αυτά τα χρήματα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Αυτό πρέπει να δούμε αν είναι θελκτικό για τράπεζες ή όχι και πώς θα μπορούσε να προσδιοριστεί και να δομηθεί το χρέος αυτό και είναι μια ε, δυνατότητα η οποία πρέπει να εξεταστεί. Πώς θα αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα σε σχέση με το ΣΥΝΑΒ και το ΒΙΝΑΒ για παράδειγμα. Πρέπει να προβληματιστούμε σε σχέση με το αυτό που προτείνετε εσείς, να επιβληθεί μία ε, λύση που, ε, που υιοθέτησαν οι ΙΠΑ. Όπως ε, είπε ο Μπράιαν, μία ολόκληρη περίοδος χρόνου, επταετής περίοδος χρειάστηκε και γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Και έχουμε κάποια εργαλεία στη διάθεσή μας, κάποια μέσα. Έχουμε για παράδειγμα την μελέτη επιπτώσεων, μελέτες επιπτώσεων. Αυτό που θα ήθελα να γίνει είναι, πρωτού αποφασίσουμε ότι δεν θα, γι... δεν θα αναλάβουμε ένα τέτοιο υψηλό κίνδυνο γιατί δεν ζητούμε από ένα αμερόληπτο όργανο να συντάξει μια σωστή πλήρη μελέτη επιπτώσεων. Ίσως αυτό μπορεί να καθυστερήσει την υπόθεση αλλά δεν κάνουμε λόγο για μια σοβαρή καθυστέρηση. Θα μπορούσε επίσης ε, να ζητηθεί να τεθεί μια εύλογη προθεσμία για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη επιπτώσεων. Θα έχουμε μια αντικειμενική όμως μελέτη επιπτώσεων επί τις οποίες θα μπορούμε να συζητήσουμε με αντικειμενικά επιχειρήματα. Συνολικά θα έδινε μια ουδέτερη αμερόληπτη αξιολόγηση επιπτώσεων και κινδύνων για το τι θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί βραχυπρόθεσμα από πλευρά μα. Αυτό που ζητώ λοιπόν ε, απλά είναι να δούμε ποιε είναι οι εναλλακτικέ λύσει και δυνατότητε. Ποιε είναι οι εναλλακτικέ ε, ε, δυνατότητε που σκιαγραφεί μια τέτοια μελέτη επιπτώσεων να δούμε την εξίσωση ε, σε σχέση με το δημόσιο χρέος, ε, τις δυνατότητες που θα έχουμε να ανταποκριθούμε. Κανείς από μας δεν γνωρίζει τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν ζητούμε λοιπόν να συνταχθεί μια μελέτη επιπτώσεων ώστε όταν επανέλθουμε να γνωρίζουμε σε μεγαλύτερο βάθος με αντικειμενικά στοιχεία το που βρισκόμαστε και τότε να συζητήσουμε για να ληφθεί μια απόφαση. Ευχαριστώ. Can I, Sorry. My ε, ε, ε, έκανα, θέλω να υποστηρίξω την πρόταση που, την, πρόταση που έκανε ο κύριος Καμάλ. Αυτό μας λέτε, έτσι, ωραία. Δεν μπορούμε να πάρουμε καμία απόφαση αυτή τη στιγμή. Απλώς για τα πρακτικά θέλετε να καταγραφεί. Πολύ ωραία. Γεια σας, φιλελεύθερη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εφόσον ε, έχετε περιορίσει το χρόνο ομιλίας μας, ε, θα ασχοληθώ με το βασικό ζήτημα, ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε το συστημικό κίνδυνο και τη μαζική αποπληρωμή των τίτλων, καθώς και το θέμα των σταθερών ΚΑΕ. Από ό,τι φαίνεται μπορεί να προκύψει συνένεση σε σχέση με τα όρια για την εξαγορά, αλλά έχει εξαφανιστεί αυτό από την πρόταση. Προτείνεται δε μια ουσιαστικότητα διαλλαγή του τοπίου των χρηματαγορών και, και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγορών. Παρότι εάν μετατραπούν ε, μαζικά οι σταθερές ΕΚΑΕ σε σταθερές δημοσίου χρέους, ε, είναι δύσκολο να προβλεφθεί αυτό ποιες επιπτώσεις θα έχει. Μπορούμε τουλάχιστον να κάνουμε κάποιες αναλογίες ε, και να δούμε ποιες διαφορές έχει το αμερικανικό σύστημα με το ευρωπαϊκό σύστημα Υπάρχουν 28 διαφορετικές εκδοχές ε, του δημοσίου χρέους ε, και έχω την εντύπωση ότι είναι ε, ούτως ή άλλως κατακαιρματισμένο το τοπίο και θα περάσουμε και λάθος μήνυμα στα κράτη-μέλη, θα τα ενθαρρύνουμε σε σχέση με το χρέος οι χρηματαγορές συνεχίζουν να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Αυτό είναι ένα δεδομένο, αλλά τώρα το να χρηματοδοτούν το δημόσιο χρέος αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Φαίνεται ότι αυτό αντιβαίνει και στο στόχο που έχουμε να βασιζόμαστε περισσότερο σε χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα και όχι σε δημόσιο χρέος. Τώρα, το πόσες σταθερές ΕΚΑΕ θα μπέσουν στον ορισμό και θα χρειαστεί να μετατραπούν σε σταθερές καί δημοσίου χρέους. Γιατί μην ξεχνάτε δεν μιλάμε μόνο για ευρώ αλλά και για δολάρια, είπα και για λίρες. Ε, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ε, τώρα η μετατροπή των λιανικών ΣΥΝΑΒ σε ΒΙΝΑΒ ε, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν το ισχυρίζομαι, απλώς ρωτάω. Και επανερχόμαστε στα αρχικά ερωτήματα. Οι σταθερές ΚΑΕ όντως χρειάζονται για να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Εγώ θα ήθελα να μην βρεθώ εμπόδιο, να μην σταθώ εμπόδιο στην ε, νομοθεσία για τα αμοιβαία κεφάλαια, όμως επειδή θα προκύψουν πολύ ριζικές αλλαγές στις ε, χρηματαγορές, θα χρειαστεί να έχουμε ξεκάθαρους στόχους. Ο στόχος δεν είναι να παρεμποδίσουμε, ξαναλέω, τη μεταρρύθμιση, αλλά να έχουμε ρεαλιστικές, βιώσιμες λύσεις τόσο για τις σταθερές όσο για τις μεταβλητές ε, ΚΑΕ. E, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την Ίνα για τη σκληρή της δουλειά. Ξέρω ότι είναι πολύ περίπλοκο να καταλήξει κάποιος σε συμβιβασμό για μια τόσο δύσκολη πρόταση. Για μας όμως από πλευράς ΓΚΟΕ η ουσία είναι τι πρέπει να γίνει. Θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτούμε και κάτι αντίστοιχο ε, της προηγούμενης έκθεσης που είχαμε στην προηγούμενη θητεία, ε, και μια γενική παρατήρηση μόνο, γιατί ακούω διάφορα εδώ. Γίνεται όλη η συζήτηση για την Ένωση της Κεφαλαίου Αγοράς και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για ε, δανεισμό εκτός τραπεζών, αλλά το βασικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο παραδοσιακός τραπεζικός δανεισμός και κανείς μέχρι τούδε δεν με έχει πείσει ότι θα πρέπει να υπάρχει μη τραπεζικός δανεισμός, ότι επειδή υπάρχει πρόβλημα με τον τραπεζικό δανεισμό θα πρέπει να αυξήσουμε το μη τραπεζικό δανεισμό για να βελτιώσουμε τις μακροοικονομικές συνθήκες. Τώρα, για αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Νομίζω ότι αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι η λιανική κατηγορία των ε, σταθερών ΚΑΕ ε, είναι σαν να ανοίγουμε τη Wall Street ε, στην ελληνική αγορά. Δεν το θέλουμε αυτό γιατί οι σταθερές ΚΑΕ είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Ε, παριστάνουν ότι είναι ουσιαστικά ρευστό ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι τέτοιο. Δεν είναι δάνεια ε, και ε, ουσιαστικά θα γίνει φορολογική βελτιστοποίηση των σταθερών ΚΑΕ και εμείς δεν το θέλουμε αυτό σε καμία περίπτωση. Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί στον κανονισμό για τα ε, κυβερνητικά σταθερά ΚΑΕ λέμε ότι θα πρέπει να είμαστε μέχρι το 3% ενώ να λέμε τουλάχιστον 3% και το ίδιο να ισχύει και για επενδύσεις σε κρατικά ομέληχα, ε, όχι μέχρι, ε, αλλά τουλάχιστον το συγκεκριμένο ποσοστό. Το ίδιο ισχύει και για τη στάθμιση του κινδύνου. Αντί των αποθεματικών και επίσης ε, διαφωνούμε για όλη αυτή τη συζήτηση με τα τέλη και τις ε, ε, Gates γιατί θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν επιλύουν το πρόβλημα αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε πανικό. Επίσης, ε, μακροπρόθεσμα ναι, όντως ε, ε, υπάρχει πρόταση για απαγόρευση εξωτερική στήριξη και εμεί είμαστε υπέρ αυτών. Δεν καταλαβαίνουμε με ποια λογική θα είναι λιγότερο ο κίνδυνο αν κοινοποιηθούν και βελτιωθούν. Υπάρχει κάποια πρόταση για βελτίωση τη διαφάνεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι να μην υπάρχει διαφάνεια, αλλά να μην συμβαίνουν κάποια πράγματα. Επίσης, ε, τα παράγωγα OTC έχουν ε, ε, αφαιρεθεί και αυτό το υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα για τους πρασίνους η Ευαζολή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την συγγήτρια για το σχέδιό της. Ε, συμφωνούμε με κάποια από τα στοιχεία της πρότασή τη, όμως ε, σε κάποια από τα βασικά ζητήματα έχουμε βασική διάσταση απόψεων. Θεωρούμε, παραδείγματος χάρη, ότι αποδυναμώνεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις σταθερές ΚΑΕ. Παρότι θεωρητικά περιορίζονται σε δύο κατηγορίες. οι σταθερέ ΚΑΕ, έχουμε σοβαρές ανησυχίες ε, ότι η παρατεταμένη προθεσμία για τις ε, σταθερές ΕΚΑΕ δημοσίου χρέους το 2020 δηλαδή και χωρίς κανένα περιορισμό στο ενδιάμεσο διάστημα αυτό θα επιτρέψει ουσιαστικά διατήρηση του μοντέλου των σταθερών ΚΑΕ για μια σειρά ετών τουλάχιστον ε, το πνεύμα της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν τέτοιο ώστε ή ε, οποιοδήποτε περιορισμό να συνοδεύεται από νομοθετική ρυθμίση ούτως ώστε στην εσωτερική αγορά να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, ένα ελάχιστο αποθεματικό ασφαλείας τουλάχιστον 3% για τις σταθερές ε, ΚΑΕ ε, και απέτηση μόχλευση σε σχέση με την οδηγία για τι κεφαλαιακές απαιτήσει καταλείται στην πρόταση της ε, εισηγήτριας ε, διότι παρατείνεται την προθεσμία μέχρι το 2020 και το αποθεματικό εισφαλείας φτάνει μέχρι το 30% αλλά για τα ε, στοιχεία με σταθμισμένο κίνδυνο ενώ ξέρουμε παραδείγματο χάρη ότι τα ομόλογα δημοσίου έχουν μηδενικό σταθμισμένο κίνδυνο άρα δεν καλύπτονται και το αποθεματικό πάει μέχρι το 3% του σταθμισμένου ε, κινδύνου το, των χαρτοφυλακίων, ε, των ε, αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς ε, και άρα αποδυναμώνεται σε μεγάλο βαθμό η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ζητούμε από την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν τους επόμενους έξι μήνες ε, να εξελογήσει τις επιπτώσεις των διαφόρων μοντέλων που καταθέτει η συγκητρία διότι πιστεύουμε πως εάν εφαρμοστούν προτάσεις της συγκητρίας της Επιτροπής μας θα διατηρηθεί το στάτο quo. Πέραν αυτού Βάσει της πρότασης της εισηγήτριας, ε, οι σταθερές ΚΑΕ δεν χρειάζονται αποθεματικό ασφάλειας ε, και άρα ε, θα είναι δυσανάλογα μεγάλος ο κίνδυνος για τους ελληνικούς επενδυτές. Ξέρουμε ότι το θέμα των, καθαρών, των σταθερών ΚΑΕ και του αποθεματικού είναι πολύ αμφιλεγόμενα ζητήματα, όμως δεν μπορούμε ε, με 7 χρόνια μετά την κρίση να πιστεύουμε ότι χωρίς ε, το αντίστοιχο τίμημα ε, θα μπορέσουμε να την γλιτώσουμε και να μετακυλήσουμε τον κίνδυνο στους επενδυτές και στους καταναλωτές. Εμείς αντίθετα είμαστε υπέρ της ενίσχυσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουμε μια μεταβατική περίοδο για την ε, μετατροπή των ε, σταθερών ΚΑΕ σε μεταβλητές ΚΑΕ. Οι μόνες σταθερές ΚΑΕ που θέλουμε να μπέσουν στην κατηγορία είναι αυτές ε, που επενδύουν σε δημόσιο χρέος, όμως με επιπρόσθετες απαιτήσει όπως ε, τραπεζική άδεια, παραδείγματος χάρη, ή ένα αντικυκλικό αποθεματικό ασφαλείας. Ε, σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις, θα συμφωνήσουμε για την κατάργηση της εξωτερικής στήριξης. Επίσης, συμφωνούμε με τους περιορισμούς για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, ε, τα πρότυπα ε, ανάκαμψης που συνάδουν όμως με την οδηγία για τις κεφαλαιοχικές απαιτήσει ε, και ξαναλέμε ότι θέλουμε να ενισχυθεί περαιτέρω η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πρώτον προβλέποντας ότι τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγορών που βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί ο εποπτικός ρόλος, ώστε τα σημαντικά αμοιβαία κεφάλαια να υπάγονται απευθείας στον έλεγχο της ΕΣΜΑ σε περίπτωση ύπαρξη σοβαρού συστημικού κινδύνου. Επίσης, ε, θέλουμε η τέταρτη οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσει ε, διακόπτει ο Πρόεδρος. Δεν μπορώ να σας δώσω άλλο χρόνο. Είστε οι μόνοι που μιλήσατε πέντε λεπτά, κυρία Ζολή. Ε, Θα σταματήσω εδώ, αλλά... Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Πρώτη Πεβάνς Μπερές. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την εισηγήτρια διότι όταν ε, κάποιος έχει βρεθεί σε ένα διέξοδο πρέπει να ε, κινηθεί, να μετακινηθεί αλλά όχι υπό οποιοδήποτε προϋποθέσεις και γι' αυτό το λόγο έχουμε ε, εμπλακεί και έχουμε ε, καταλήξει ένα τέλμα διότι ε, υπάρχει ανισότιμη κατανομή των χρηματαγορών ε, στα κράτη-μέλη και αυτό το βλέπουμε και συζητήσει στο Συμβούλιο και γίνεται μια αξιολόγηση βάσει τριών κριτηρίων που μας προτείνει η συγκήτριά μας και έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν θα τα πάρουμε την ίδια σειρά διότι το πρώτο κριτήριο είναι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η συστημική κίνδυνη. Ωραία. Δεύτερο κριτήριο ο τρόπος με τον οποίο η χρηματαγορά μπορεί ναι ή όχι να διευκολύνει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και τρίτο κριτήριο, κριτήριο με ποιο τρόπο ε, χρησιμοποιούμε σε περίπτωση ατυχήματος τα χρήματα του φορολογουμένου. Ε, βλέποντας αυτά τα τρία κριτήρια, ως Ευρωπαίοι νομοθετές θα καλούμαστε να βρούμε την σωστή ισορροπία και όχι να υποκύψουμε στο συντηρητισμό κάποιων κλάδων ή κάποιων ε, νομομαθών ε, ενός οργανισμού χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που ε, μπορεί να ισχύει από νομικής άποψης αλλά δεν εξυπηρετεί αυτά τα τρία κριτήρια που προανέφερα. Να μην ε, προσφεύγουμε δηλαδή στα χρήματα των φορολογουμένων, ε, να βρούμε έναν ισορροπημένο τρόπο να χρηματοδοτούμε την οικονομία και να διασφαλίσουμε τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Λοιπόν, ως προς τη διαφοροποίηση, δεν χρειάζεται τώρα να μακρηγορήσω γι' αυτό γιατί το αναγνώρισε και η διασηγήτρια και το είπαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, το να παίρνουμε ένα κομματάκι από τη μία πρόταση, το αμερικανικό μοντέλο δηλαδή, και να το συνδυάσουμε με τα δικά μας, ε, παρουσιάζει μια διπλή δυσκολία. Πρώτον, ε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον τρόπο λειτουργίας ε, των σταθερών ΚΑΕ και πώς ακριβώς χειρίζονται το χαρτοφυλάκιό τους ως προς το δημόσιο χρέος, διότι δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, διότι έχουμε πάρει ένα μόνο κομμάτι της πρότασης. Ε, τώρα, με ανησυχούν δύο πράγματα. Πρώτον, τι γίνεται με την ε, περιβόητη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αποθεματικό ασφάλειας. Ε, νομίζω ότι είναι στον πυρήνα του προτινόμενου συστήματος, ε, διότι Μόνο έτσι οι σταθερές ε, ΚΑΕ μπορούν ε, να ανταποκριθούν ε, στις προσδοκίες όλων που προέκυψαν από την κρίση και δεύτερον με τη διαφοροποίηση των σταθερών ΚΑΕ προς το δημόσιο χρέος δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς θα χρηματοδοτήσουμε την πραγματική οικονομία. Για μένα παραμένει ακύρωτο το μυστήριο, δεν μου έχει δοθεί καμία απάντηση. Θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να μου το εξηγήσετε. Ευχαριστώ Σβεν Γκίγκολτ είμαι πολύ σύντομος. Πρέπει να πω, δεν θέλω να επισέλθω σε βάθος στην ουσία του θέματος. Η ερώτηση κλειδί είναι, τα ταμεία θα έπρεπε να έχουν την ίδια λειτουργία όπως οι τράπεζες. Αυτό είναι ο πυρήνας της συζήτησης. Πολλά επιχειρήματα ακούστηκαν για την προστασία κάποιων πρωτήτων επιχειρησιακών αν αυτό θα είχε μεγάλες ή όχι επιπτώσεις κτλ. Εγώ είμαι πεισμένος για το ότι αν εγγυόμαστε μια συγκεκριμένη αξία είναι τότε κάποιος τράπεζα και αν είναι κάποιος ταμείο πρέπει να έχει κειμενόμενη αξία. Εκτός αν κάποιος τρίτος αναλαμβάνει αυτόν τον κίνδυνο. Δεν μπορεί απλά να είναι κάποιος σύναυ και έτσι να είναι υποχρεω, υποχρεωμένος να, να υπόκειται σε κυκλικές δράσεις. Πολλοί από τους ομιλητές δεν αναφέρθηκαν στα στοιχεία και αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε ήδη. Έχουμε μία έκθεση του Ευρωπαϊκού ε, ε, Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και είναι σαφή, σαφή τα συμπεράσματα θα έπρεπε για μακροοικονομικούς ε, λόγους ε, να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτή την κυκλική ε, σύσταση κινδύνων. Και εδώ ζητούν κάποιοι νέα μελέτη επιπτώσεων. Ως συντονιστής μπορώ να πω ότι είναι προφανές που θα οδηγήσει κάτι τέτοιο. Θα σήμαινε ότι περνάμε στη Λουξεμβούργια Προεδρία και αυτό θα τέριαζε πολύ καλά με ένα Ιρλανδό εισηγητή, ένα Βρετανό εισηγητή και έναν άλλο Βρετανό σκιώδη εισηγητή και τα λοιπά και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Και θέλω ανοιχτά να σας πω πώς το βλέπω και εσείς μπορείτε επιθετικά ίσως να αντιδράσετε. Αλλά θέλω να σας πω σε μια ανοιχτή συζήτηση ότι εγώ ανησυχώ για το κύρος και την αξιοπιστία αυτής της κοινοβουλευτικής επιτροπής. Κατά παρελθόν είχαμε πολύ ευε, μεγάλες ευαισθησίες. Δεν ε, έπαιρνε κάποιος μια εισήγηση μια έκθεση αν υπήρχε η εντύπωση ότι θα υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά κάποια συγκεκριμένη χώρα. Τώρα έχουμε μια συμπίκνωση ε, σε συγκεκριμένα θέματα συγκεκριμένων ευρωβουλευτών και αυτό δεν είναι θετικό. Έχουμε κίνδυνο που αναφύεται να αποδυναμωθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Επιτροπή μας. Το έχουμε εδώ σε αυτή την περίπτωση και με την ε, μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα. Και έτσι δεν έχουμε έχουμε αντιδράσει όπως θα έπρεπε όσον αφορά την αποδυνάμωση. Ε, βρίσκω ένα κίνδυνο το Ευρωκοινοβούλιο να παρεκκλίνει από την παράδοσή του να ενισχύει την χρηματοοικονομική σταθερότητα όταν είχαμε έναν επίτροπο κατ' παρελθόν τον Ιρλανδό Μαγκρίβι να αποδυναμωθούν οι διατάξεις όσον αφορά τις πτυχές της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ αρνητικό και αυτό φαίνεται ότι είναι η κατεύθυνση στην οποία πορευόμαστε και μπορώ και περισσότερα στοιχεία να αναφέρω βλέποντας το τι γίνεται με τις λεπτομέρειες όσον αφορά τις κεφαλαιακές αγορές. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να είμαστε πολύ σοβαροί όσον αφορά τις προσδοκίες των πολιτών να είμαστε αυστηροί όσον αφορά τις ε, διατάξεις ε, για την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Να μην αποδυναμώσουμε τα πράγματα γιατί θα είναι κίνδυνο. Μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων, ο κύριος Φων Βάιτζάκερ, ε, νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω με τι χρηθεί η Λίνα και τι έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό το τόσο δύσκολο θέμα. Πρόκειται για ένα από αυτά τα θέματα όπου όλοι προσπαθούν να σου πούνε ότι μπορείς να έχεις και την πίτα ολόκληρο και το σκύλο χορτάτο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν γίνεται ή θα διατηρήσουμε τον τομέα των σταθερών ΚΑΕ που είναι ένας μεγάλος τομέας και το γνωρίζουμε όλοι και δεν θα αντιμετωπίσουμε το συστημικό κίνδυνο που εμπεριέχει ή θα πρέπει να πούμε και να σταματήσουμε να υποκρινόμαστε ότι οι σταθερές ΚΑΕ είναι πολύ καλό κεφάλαιο. Ε, πρέπει να κάνουμε μια επιλογή και θα πρέπει να αποφασίσουμε. Αν υπάρχει μια ερώτηση που πραγματικά αν θέλουμε να κάνουμε μια αξιολόγηση θα έπρεπε να κάνουμε, που εγώ δεν θεωρώ ότι χρειάζεται, ε, είναι πολύ απλή ερώτηση. Τι η προτινόμενη νομοθεσία και η κατάσταση που αποτίθεται ότι θα επιλύσουν οι σταθερές ΚΑΕ που ε, έχουν τεράστιο συνδυμικό κίνδυνο λόγω των ε, υφερπόντων και όχι τόσο κρυφών ε, ε, κεφαλαίων στοιχείων ενεργητικού που ε, εκμεταλλεύονται σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Αυτή είναι η μόνη ερώτηση που θα έπρεπε να τεθεί και πραγματικά θα με ανησυχούσε ιδιαίτερα εάν η απάντηση στην ερώτηση είναι ότι αυτό το αποθεματικό ασφαλείας του 3% θα διαχυθεί ακόμα περισσότερο. Οι σταθερές ΚΑΕ, οι οποίες ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο προκέπκυψαν και διαχύθηκαν αυτά τα προβλήματα της Lehman Brothers, ε, νομίζω ότι μας κάνει την ερώτησή μας πολύ απλή. Στο παρελθόν δεν τα καταφέραμε και αν συνεχίσουμε έτσι ούτε θα τα καταφέρουμε τώρα και κατά πάσα πιθανότητα, όχι για τους ίδιους λόγους που λέει ο Σβέν, αλλά θα γίνουμε περίγελος οποιοδήποτε πραγματικά ρίξει μια σοβαρή ματιά στους συστημικούς κινδύνους που ολοχεύουν. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τελευταίο ο πριν δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Σιλβί Γκουλάρ. Ευχαριστώ πολύ. Σβέν, χαίρομαι όταν κάνεις συνδέσει Τον παλιό καλό καιρό της παλιάς θητείας θυμόμουν ότι είχαμε μόνο Γερμανούς εισηγητέ στο θέμα αυτό, το Deposit Guarantee Scheme για παράδειγμα. Πρέπει πάντα να αποφεύγουμε να υπάρχουν κάποια εθνικά ε, συμφέροντα είτε στο θέμα αυτό είτε στο άλλο και δεν θέλουμε εδώ να κατηγορήσουμε τους συναδέλφους. Νομίζω ότι οι φιλελεύθεροι έκαναν την καλύτερη δυνατή επιλογή και το μόνο που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε κι εσείς. Τώρα, σοβαρά. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και εμένα με ανησυχούν δύο πράγματα στην πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας. Πρώτον, ε, η αλλαγή σε σχέση με αυτό που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν χρειάζεται μελέτη επιπτώσεων, αν πρέπει να ρωτήσουμε την άποψη της e SRB και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά όταν αλλάζει τόσο η λογική νοκειμένου, τότε σίγουρα θα πρέπει να θέσουμε ερωτηματικά και ε, η διαφορά σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να τους ακολουθήσουμε κατά πόδας. Ε, δεν είναι θέμα αν είναι καλές ή όχι πρακτικές της, των ΗΠΑ, δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά αν οι πρακτικές της δικής μας οικονομίας είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση του θέματος κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Λίντερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους βουλευτές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και εις βάθος συζήτηση που γίνεται. Είναι δύσκολο το ζήτημα και νομίζω βρεθήκατε ήδη στον πυρήνα της πρότασής μας, ε, δηλαδή ε, με ποιο τρόπο μπορεί να παραμείνουν βιώσιμες οι χρηματαγορές. Μετά από μακροσκελέστατες συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο, διαπιστώνουμε ότι διείστανται απόψε μεγάλο βαθμό μάλιστα και ε, γι' αυτό ε, η συγγήτρια και άλλοι βουλευτές προτείνουν συμβαστικές λύσεις οι οποίες συζητούνται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο το ζήτημα και όπως είπατε, ο αντίκτυπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση είναι πολύ καλός και λεπτομερής. Εάν υπάρχουν άλλα ζητήματα που θέλετε να μελετήσουμε, μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη δυνατότητα να σας βοηθήσουμε να ερευνήσετε διεξοδικότερα κάποια ζητήματα. Για το χρονοδιάγραμμα φυσικά έχουμε διεθνείς υποχρεώσεις ε, τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούμε και ξέρουμε ότι χρειάζεται πολλούς χρόνος για τη διεξαγωγή μελέτης αντικτύπου. Πάντως, αν χρειάζεστε τεχνικές συμβουλές, είμαστε στη διάθεσή σας και περιμένουμε το αποτέλεσμα των συζητήσεων της εισηγήτριας με τους σκιώδεις ε, για το μέλλον των σημαστικών λύσεων παθή. Thank you to the Commission. Ευχαριστούμε την, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είστε διαθέσιμος λέτε για μας βοηθήσετε, αλλά δεν σας το ζητήσαμε ακόμη, είστε πολύ γρήγορος. ο κύριος Γκίγκολ, ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατάλαβα καλά αυτά που είπατε. Δεν υπερασπίζεστε πλήρως την πρότασή σας. Απάντηση. Όταν υποβάλαμε την πρόταση θεωρούσαμε ότι ήταν η καλύτερη το αμερικανικό μοντέλο, αν μεταφερθεί αυτούσιο στην Ευρώπη, θα, λόγω διαρθρωτικών ε, ε, διαφορών θα δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα. Και γι' αυτό εμείς προτείναμε τη λύση του αποθεματικού ασφαλείας. Λοιπόν, είναι καλή πρόταση, αλλά ταυτόχρονα έχουμε επίγνωση του ότι έχει μπει το θέμα σε μια πολιτική διαδικασία και παρότι εξακολουθούμε να την υπερασπιζόμαστε, θέλουμε να φανούμε και επικοδομητικοί. So apparently the answer to your question is... Ναι, δηλαδή κύριε Γίγκολ, τα πάντα ή μάλλον εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ερώτημά σας. Εισήγητρια, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Κάποιοι μου είπανε τι αμαρτίες πληρώνεις Νίνα και σου έλαχε αυτός ο φάκελος. Ε, κοιτάξτε, προσπαθώ να βρω έναν τρόπο για να προχωρήσουμε. Είμαι, σίγουρα δεν είναι τέλεια η πρότασή μου. Είδατε στην πρόταση ότι υπάρχει σαφής ε, διαφοροποίηση και δυσκολευόμαστε να βρούμε τη μέση οδό. Προσπαθούμε όμως, προσπαθούμε να καταλήξουμε σε ένα πακέτο διότι στο κάτω-κάτω της γραφής το σημαντικό είναι να έχουμε κάτι. Και ξεκάθαρα προκύπτει και αυτό και από την προηγούμενη και από τη σημερινή συζήτηση ότι αυτός είναι ο λόγος, η διαφορά απόψεων δηλαδή, για τον οποίο δεν έχουμε καταλήξει ήδη σε λύση. Δηλαδή, οι σκιώδεις ε, πρέπει να έρθουν να συναντηθούμε, να όχι να υπερασπιστούν και να εμένουν στις θέσεις τους όλοι, αλλά να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια συμβαστική λύση. Ε, τώρα λένε κάποιοι ότι αντιγράφουμε το αμερικανικό μοντέλο. Με την ναι, SEC τι έγινε, έκανα μία συζήτηση μόνο περιορισμένη κιόλα και με τους, ε, μίλησα με τόσους διαφορετικούς ε, φορείς για να βρούμε μία διέξοδο, για να διαχειριστούμε τον κίνδυνο με τον ενδεδειγμένο τρόπο όπως σωστά το έθεσε ο Μπράιεν. Προσπαθώ λοιπόν και εγώ να βρω τρόπους για να διαχειριστούμε τον κίνδυνο, γιατί έτσι μπορούν να παραμείνουν όσοι έχουν σταθερές ΚαΕ. η Επιτροπή ε, έχει εξετάσει όλα αυτά τα εναλλακτικά σενάρια. Αυτή είναι μία εκδοχή, ένα σενάριο και αυτό ε, καταθέτω. Έχουμε το χρόνο 2020, αυτό δεν το κάνουν ε, στις ΗΠΑ. Δεν πρόκειται τώρα να κάτσω να σας πω σε ποια σημεία διαφέρει δική μου πρόταση από το αμερικανικό μοντέλο μπορούμε να κάνουμε ένα μείγμα, λέμε Α, δεν θέλουμε το αμερικανικό μοντέλο. Ε, λέτε εσεί ότι εκείνοι το συζητάνε έξι χρόνια και εμεί πέντε χρόνια το συζητάμε. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Ε, από την εμπειρία που έχουμε από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία στην οποία δεν καταλήξαμε σε συμφωνία βλέπουμε ότι παραμένει η κατάσταση και άρα τι αλλάζει να περιμένουμε άλλους λίγους μήνες, άλλους λίγα χρόνια, τι αλλάζει. Το σημαντικό είναι τι συμβαίνει τώρα διότι ε, συμφωνώ, διαφωνώ με πολλά από αυτά που λέει ο Σβέν, αλλά συμφωνώ με αυτό που λέει ότι ε, διακυβεύεται η αξιοπιστία μας. Δεν είμαστε το Συμβούλιο. Γιατί συζητάμε σαν να είμαστε το Συμβούλιο. Δεν είμαστε η Επιτροπή. Ε, η δική μας η δουλειά είναι να ελέγχει, να εξετάζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι οι ιερές για μας οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να ακέρες να τις υιοθετούμε. Δεν είναι ο ρόλος μας. Άλλαξαν και τα δεδομένα εντωμεταξύ σε ορισμένου τομεί, ε, Ζητάνε κάποιοι νέα αξιολόγηση αντικτύπου. Μα όλα αυτά τα νούμερα που σας έδωσα ε, απορρέουν από την αξιολόγηση αντικτύπου που έγινε το Σεπτέμβριο του 2013 από τη Στατιστική Υπηρεσία. Τι αλλάζει, εν πάση περιπτώσει. γιατί ζητάμε νέα αξιολόγηση αντικτύπου. Μιλάμε για τα ποσά που ισχύουν για τον δημόσιο τομέα, τα ανώτερα όρια, έχουμε τα δεδομένα για το λιανικό για τις λιανικές επενδύσεις δεν θα αλλάξει τίποτα ουσιαστικά και το μόνο που θα κάνουμε είναι να καθυστερήσουμε περισσότερο και κάθε φορά που κάποιος βουλευτής προκύπτει μια νέα πρόταση δεν είναι λύση να ζητάμε νέο, νέα αξιολόγηση αντικτύπου. Για φανταστείτε, αν προκύψει, αν, αν ανακύψει ένα πρόβλημα στις χρηματαγορές τους επόμενους μήνες, τι θα κάνουμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Ας δούνε όλοι με ποιο τρόπο μπορούν να συμφωνήσουμε ένα πακέτο που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Εγώ πιστεύω το σημαντικότερο είναι ε, να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται και να μην περιμένουμε την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Κάποιοι δε κάνουν ισχυρισμού ε, για το, ε, την προηγούμενη σταδιοδρομία κάποιον ε, ή για το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εκπροσωπούμε 500 εκατομμύρια πολίτες και δεν μπορεί να λέει κάποιο, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε Βρετανή εισηγήτρια, πρέπει να βάλει μεγάλο εισηγητή σε κάποιο άλλο ζήτημα, είναι Ιρλανδό ο Σκιώδη. Πρέπει να, να τα ξεπεράσουμε αυτά επιτέλου και να πούμε ε, δεν γίνεται να συνεχίσουμε με αυτό το τέλμα, με αυτό το αδιέξοδο. Πρέπει να, να εξασφαλίσουμε ότι θα φτιάξουμε ένα πακέτο που να ομαδοποιεί τις απόψεις όλων και αυτό προσπαθώ να κάνω. Ίσως δεν έχω συμπεριλάβει όλα τα ζητήματα. Είμαι πρόθυμη να συνεχίσω τις προσπάθειες. Αυτά που μας λέει ο κύριος Ντεμάς, η κυρία Ζολή, αυτά που είπε ο Μπράιεν, ο Σαΐντ και ο κύριος Ζέζεκ. Ο, ο, τους θα συνεργαστούμε και για να μην χάσουμε την αξιοπιστία μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να βιαστούμε, να βρούμε έναν τρόπο για να ε, βγούμε από αυτό το ε, αδιέξοδο την ε, Πέμπτη, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Έχουμε τώρα στις 11 Δεκεμβρίου στις 12 την προθεσμία για τις ε, τροπολογίες, 21 ε, Ιανουαρίου θα το ε, εξετάσουμε, το εξετάσουμε την έκθεση, 23-24 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε, ενδεχομένως αν λάβουμε έτοιμα για εκπόνηση νέας μελέτης αντικτύπου θα την εξετάσουν οι συντονιστές, δεν ξέρω. Εάν μπορείτε να εξετάσετε και μια εναλλακτική λύση. Αν ε, δοθούν και άλλε δύο-τρει μέρε, ε, παραταθεί η προθεσμία και την υποβολή τροπολογιών κατά τρει-τέσσερι μέρε, θα μπορούσε ενδεχομένω η συγγήτρια να βρει μια λύση, μια εναλλακτική λύση για το θέμα τη μελέτη αντικτύπου και μπορούμε να το κοινοποιήσουμε στα μέλη τη Επιτροπή στη συνέχεια. Τι λέτε, συγγήτρια. Ε, δεν, ε, πρόεδρε, σε δύο-τρει μέρε τέτοια απόφαση δεν μπορούμε να λάβουμε. Έχουμε πρόγραμμα και έχουμε πολλά άλλα νομοθετήματα δεν είναι εύκολο τώρα να καθυστερήσουμε και να παρατείνετε τις προθεσμίες. Ε, δεν γίνεται απλώς να, χώσετε την έκθεση ε, όπου, όπου μας βολεύει εμάς. Όχι, όχι, λέει ο Πρόεδρος, ε, θα, παραμείνει το χρονοδιάγραμμα όσο έχει και η ψηφοφορία και η εξέταση κτλ. Απλώς Ρώτησα εάν παραταθεί μόνο η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών κατά δύο-τρει μέρε, μα βοηθήσει. Η συγγήτρια, ναι, ναι, ναι, αλλά άμα δεν αλλάξει συνολικά το χρονοδιάγραμμα, κανένα πρόβλημα. Την επόμενη Τετάρτη, δηλαδή, στο Στρασβούργο, λίγε μέρε παραπάνω. Ε, μία ερώτηση. Από ό,τι κατάλαβα, οι συντονιστέ ε, θα δουν το θέμα να εξετάσουν το θέμα ε, της εκπόνησης νέας μελέτης αντικτύπου. Απάντηση του Πρόεδρου είναι αν μόνο υποβληθεί το αίτημα επισήμως. Ωραία. Ε, αυτό σημαίνει ότι διατηρείται το φυστάμενο χρονοδιάγραμμα για την πρόταση απάντηση ναι, ναι, ναι και ε, μια ε, ίσον σημασία αλλαγή γίνεται για την προθεσμία υποβολής τροπολογιών κατά λίγες ημέρες. Φυσικά οι συντονιστές αν το επιθυμούν μπορούν να επανέλθουν στο ζήτημα να συζητήσουν την πρόταση εάν κατατεθεί η πρόταση, ξαναλέω, για εικόνες νέας μελέτης. Διατηρείται το χρονοδιάγραμμα και παρατείνεται η προθεσμία. Επαναλαμβάνω, 17 Δεκεμβρίου για τις τροπολογίες, 21 Ιανουαρίου εξέταση των τροπολογιών, 22-23 Φεβρουαρίου ψεφοφορία στην ΕΚΟΝ και ε, η δεύτερη ε, ολομέλεια του Μαρτίου. Ενδεικτικό αυτό, έτσι. Point of our agenda. Σημείο 7, τελευταίο κιόλας. Ε, ζητώ συγγνώμη από την εισηγήτρια. Προσπάθησα να τηρήσουμε την προθεσμία. Θα περάσουμε στους δείκτες Κόρα, σου δίνω ε, το λόγο. Ευχαριστώ πρώτα. Ξεκινώ με πολλές ευχαριστίες προς τους σκιώδεις εισήγητες για την ευκαιρία να έχουμε ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα ως χαρτοφυλάκιο. Πρωτού περάσω στην ουσία θέλω να, α, να περάσω να διεξέλθω κάποια διοικητικά θέματα. Προσπαθώ το σχέδιο έκθεσης να ολοκληρωθεί κατά τα τέλη αυτής της εβδομάδας. Και υποθέτω ότι θα δημοσιευθεί κατά το πρώτο ήμιση της επόμενης εβδομάδας. Και επίσης το τελικό κείμενο της έκθεσης υπάρχει στην ιστοσελίδα μου διαθέσιμο και ο κατάλογος όλων των οργανώσεων που είχα επαφές για τις βέλτιστες πρακτικές benchmarks θα δημοσιευθεί και θα δημοσιοποιηθεί επίσης όποιος ενδιαφέρεται θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία προσπαθώ να παραμείνω πιστή στο χρονοδιάγραμμα με προθεσμία για τις τροπολογίες για την 20η Ιανουαρίου 2015. Περνάω στα θέματα ουσίας του σχεδίου έκθεσης. Όπως προανέφερα, είναι ένα ευρύτατο και πολυσύνθετο χαρτοφυλάκιο. Μια γενική προσέγγιση λοιπόν και επικέντρωση των κυριότερων θεμάτων του σχεδίου έκθεσης. Η γενική μου προσέγγιση για πρόσθετη νομοθεσία, περαιτέρω νομοθεσία, ώστε να αποφευθούν οι χειραγωγήσεις ε, των προδιαγραφών. Και έχει αυτό με την ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Οι προδιαγραφές ε, benchmarks είναι πάρα πολύ σημαντικές για την αξιόπιστη λειτουργία των χρηματιστηριακών αγορών, των αγορών αγαθών κτλ. Και αυτό όσον αφορά την αξιοπιστία των benchmarks καθώς επίσης και την ε, ε, μη λειτουργική ε, πτυχή αυτών των στοιχείων που θα μπορούσαν να είχαν αρνητική επίπτωση στις αγορές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα benchmarks. Οι χρηματιστηριακές αγορές και η ευρύτερη οικονομία εξυπηρετούνται καλύτερα από τέτοιες προδιαγραφές που παράγονται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο. Από αυτά τα σκεπτικά απορρέουν οι ανάγκες πρώτων. Να δώσουμε την δυνατότητα στους χρήστες των benchmarks δίνοντάς τους περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την εκπόνηση αυτών των στοιχείων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν καλύτερα τις αποφάσεις όσον αφορά τη χρήση τους και επιβάλλοντας πειθαρχία στην αγορά διοικητικά. Δεύτερον, να εφαρμόσετε σαφώς η αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά ε, ε, την επιβολή διατάξεων ώστε benchmarks με συστημική σπουδαιότητα να υποβάλλονται σε πιο αυστηρές διαδικασίες και διεργασίες ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει η ευρύτερη διάθεση αυτών των στοιχείων σε εύλογες τιμές για τους χρήστες για την αναλογικότητα και τη διαφάνεια για κέρια σημασία benchmarks δηλαδή με πολύ μεγάλη αξίας ή ε, συστημική αξία αυτών των δεδομένων είναι σημαντικό να υπάρχουν δεσμευτικές προδιαγραφές και με βάση διεθνείς αρχές που θα έχουν συμφωνηθεί. Αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν μια αναλογικότητα όσον αφορά την υιοθέτησή τους καθώς επίσης και τη χρήση τους για τέτοιου είδους benchmarks που δεν θα έχουν αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει όμως να έχουν παρόλα αυτά μεγάλη ευρύτερη διαφάνεια για τους χρήστες και τελικούς χρήστες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί απαιτώντα από τους διαχειριστές να δημοσιοποιούν δηλώσεις αξιοπιστίας για αυτές τις benchmarks με πιστοποίηση ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών καθώς επίσης και άλλων απαιτήσεων επιβάλλοντας ε, ευρύτερες ε, δεσμευτικές ε, τέτοιες διατάξεις απεριόριστα θα δημιουργούσε τον κίνδυνο να επιβληθούν περιτά κόστη. Τέτοιου είδου περιτά κόστη μπορούν να περιορίσουν τη χρήση αυτών των benchmarks και με τη μετακύληση στους τελικούς χρήστες θα περιόριζε το εύρος της χρήσης αυτών των στοιχείων από τους χρήστες σε μια συγκυρία όπου θα έπρεπε να έχει την ανώτατη προτεραιότητα η προσπελασιμότητα αυτών των στοιχείων στους χρήστες. Χρειάζονται λοιπόν αυτές οι ε, για τα αγαθά με βάση τις ε, παρεμβάσεις των, ε, των εκείνων που παράγουν αυτά τα στοιχεία που θα ευθυγραμμίζονται πάνω με τις ανάγκες το να καθορίζει κανείς τον κέριο χαρακτήρα τους που έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Διτή προσέγγιση απαιτείται. Πρώτον, benchmarks με ευρύτερα πλαίσια πάνω από 500 δις μέσα σε εύλογη περίοδο θα πρέπει να θεωρούνται κρίσιμη σημασίας. Ωστόσο, μία ποσοτικοποίηση αποκλειστικά δεν ε, ε, είναι ενδεδειγμένη για την ανάπτυξη ενός θετικού πλαισίου αγοράς. Γι' αυτό πρέπει να, ληφθούν υπόψη, ε, να ληφθεί υπόψη η ένταξη benchmarks με βάση κριτήρια που μπορούν να αξιολογήσουν τη συστημική σπουδαιότητά τους. Σε αυτό το εγχείρημα είναι σημαντικό να εφαρμοστούν οι ίδιες αρχές πανενοσιακά Γι' αυτό όπου έχουν έκθεση σε πολλαπλά κράτη-μέλη ε, τέτοια benchmarks, η τελική απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, για εθνικού, ε, ε, εθνικής χρήσης επίπεδα μπορούν τα, οι αρχές των κρατών μελών να αποφασίζουν. Για τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό benchmarks, διασφαλίζοντας την λειτουργικότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος και της πραγματικής αγοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνει λειτουργικές διατάξεις και για τρίτες ε, χώρες και εμπλεκόμενους. Αυτή τη στιγμή Καμία νομοθεσία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει θέση σε λειτουργία ένα τέτοιο ευρύτερο πλαίσιο και ούτε αναμένονται σημαντικότερες τέτοιες εξελίξεις κατά το άμεσο μέλλον. Γι' αυτό ένα καθεστώς τρίτης, ε, τρίτων χωρών ε, με ένα ε, σύστημα ισοδυναμίας δεν θα ήταν επαρκές. Ταυτόχρονα ένα πλαίσιο ισοδίκαιο θα πρέπει να διασφαλίζεται από την ΕΕ. Γι' αυτό χρειάζονται πρόσθετα μέσα και εργαλεία να διασφαλίζεται η πρόσβαση ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους σε τρίτες χώρες. Και ισοδύναμες αποφάσεις που θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες δράσεις. Η οθέτηση από διοικήσεις τρίτων χωρών και μια σωστή διαπίστευση ή αναγνώριση των ε, ε, αρχών αυτών σε σχέση με τρίτες χώρες ε, μέχρι ότου να μπορέσει ένα συνολικό πλαίσιο νομοθετικό να υιοθετηθεί και να λειτουργήσει συνολικά για αυτές τις χώρες. Μια τελική παρατήρηση, ενώ συγκρούσεις συμφερόντων ή άλλες αδυναμίες μπορεί να εντάσσονται σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σε ένα πρέπει να αναγνωρίσουμε ταυτόχρονα ότι οι, τα benchmarks που χρησιμοποιούν άλλες, άλλους δείκτες ή συνδυασμό δείκτων όπως για παράδειγμα για τις ε, επιδόσεις ε, ε, benchmarks πρέπει να θεωρούνται ένα, ένα επιπλέον πρόσθετο μέσο. Διαθέτοντας τέτοιες πληροφορίες στους χρήστες και στα θεσμικά όργανα βοηθά να διασφαλίζεται και να βελτιώνεται η διαφάνεια και λειτουργικότητα των αγορών διασφαλίζοντας στους τελικούς χρήστες καλύτερη προστασία έναντι στρεβλής χρήσης αυτών των benchmarks. Γι' αυτό εποπτευόμενοι φορείς με τις ε, διαπιστεύσεις αυτές πρέπει να καταβάλουν μια πρόσθετη προσπάθεια ώστε να ενημερώνονται οι χρήστες για τις ε, ιδιομορφίες αυτός και οι εξεχωριστές ιδιότητες αυτών των benchmarks. Νομίζω μπορώ να επαρκεστώ σε αυτές ε, τις παρατηρήσεις εισαγωγικά πρόεδρε. Και προσβλέπω και αδειμονώ στο να ακούσω τις απόψεις των συναδέφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Χοκμαρκ θα λάβει τον λόγο. Thank um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον κύριο Νίτε Μάιερ, ο οποίος ζητά συγγνώμη διότι δεν θα μπορέσει να παραστεί σήμερα. Είναι στην Κουάλα Λουμπούρ. Έχει ε, πάει για τη διάσκεψη των κεντρικών τραπεζών. Πήγε λοιπόν στην Κουάλα Λουμπούρ και μ' με να δω τον έρμο εδώ. Μπορεί να μου φέρει κανένα μπλουζάκι, δεν ξέρω μου ζητήθηκε να σας διαβιβάσω κάποιες από τις βασικές τους παρατηρήσεις που συνάδουν με τα όσα είπε μόλις η συγγήτρια. Υπάρχει μια συνεννόηση, συμφωνεί με τα όσα λέει η συγγήτρια και την ευχαριστεί. Ε, βέβαια η παραποίηση του Λίμπορ και του Γιουρουμπόρ οδήγησε σε μεγάλη ανησυχία και υπογράμμισε και τη σημασία των δικτών αναποράς. Επειδή υπάρχει ο κανονισμός και η οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς, ε, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και έχουμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Και έχουμε ταυτόχρονα και την απάντηση του G20 για την έγκριση των ε, αρχών ε, της Διεθνούς Οργάνωσης των Επιτροπών Χρηματιστηριακών Αξιών, που είναι κάτι το οποίο δέχονται οι αγορές. Ο κύριος Νίδη Μαΐερ έχει τρία θέματα τα οποία θα ήθελε να θέξει. Καταρχάς ε, την επέκταση του κανονισμού, διότι αναγνωρίζουμε ότι όσο ε, μεγαλύτερη είναι η έκτασή του, τόσο πιο εύκολο θα είναι να εφαρμοστούν και μπορεί να υπάρχει και κίνδυνος ουσιαστικής αύξησης των ε, ρυθμιστικών απαιτήσεων. Επίσης υπάρχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το καθεστώς ΑΙΟΣΚΟ και το καθεστώς των τρίτων χωρών. Όταν ε, ετοιμάστηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν σαφές τι θα γίνει σε σχέση με τις αρχές του ΑΙΟΣΚΟ. Αυτή τη στιγμή ε, λίγο πολύ αποτελούν τη βάση για τον κανονισμό στις περισσότερες χώρες και κατά πάσα πιθανότητα και ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει το νέο πρότυπο που θα μπορούμε να εφαρμόσουμε εδώ. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι υπάρχει κατάλληλη ισορροπία ε, μεταξύ των δύο. Σήμερα κάποιοι δείκτες αναφοράς χρησιμοποιούνται από αυτούς που συμμετέχουν στην αγορά, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, ε, κάνει την ίδια χρήση. Επομένως, ε, θα πρέπει οι διαχειριστές να δουν αν επαρκούν, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει περισσότερη νομοθεσία. Δεν ξέρω αν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες αναφοράς για τα ευρωπαϊκά χρήματα και αυτό μπορεί να έχει πολύ σημαντικέ συνόπειε για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και για του πολίτε. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι αν θέλουμε να θεωρήσουμε ότι οι δείκτε αναφορά στο ΕΟΣΚΟ είναι ασφαλεί και να μπορούμε να έχουμε ε, ε, ασφάλεια για του επενδυτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Ε, υπάρχει και το θέμα της διαφάνειας, το οποίο αναφέρθηκε και σήμερα εδώ. Σε γενικές γραμμές, η παρατηρήση του κυρίου Νίντεμπάιερ είναι ότι πρέπει να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού, να διευκρινίσουμε το θέμα των εκτελεστικών πράξεων, να αυξήσουμε τη διαφάνεια και ο κανονισμό να συνάδει όσο το δυνατόν περισσότερο με τι αρχέ ΑΙΟΣΚΟ και οι δείκτε αναφορέ που εφαρμόζονται θα είναι ανάλογοι με αυτού του ΑΙΟΣΚΟ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για την καλή τη δουλειά και την αμοιβαία συνεννόηση που υπάρχει και προτείνουμε οι συντονιστέ να ζητήσουν από την αρμόδια κοινοβουλευτική υπηρεσία να κάνει μια εκτίμηση των επιπτώσεων και να τη λάβει υπόψη της υπό το φως και των νέων εξελίξεων που έχουμε. Όλα αυτά από πλευράς κύριου Νίδερ Μάιερ και από μένα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για τους σοσιαλδημοκράτες. Φερνάντες Αλβάρες παρακαλώ. Καλό σας απόγευμα πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα να συγχαρώ είναι εισηγητέα. Τις τελευταίες εβδομάδες κάναμε μια έντονη σε βάθος δουλειά και εμπιστεύουμε στο ότι τις επόμενες εβδομάδες ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε το έργο ώστε να προετοιμαστεί αυτός ο κανονισμός τόσο το δυνατόν νωρίτερα. Για τις ανάγκες αυτής της ρύθμισης υπάρχουν φυσικοί λόγοι όταν υπήρξαν περιπτώσεις χειραγώγησης, περιπτώσεις που γνωρίσαμε από τον τύπο κατά τα τελευταία χρόνια αλλά και τους τελευταίους μήνες διότι η χειραγώγηση δεν ήταν μόνο θέμα Euribor ή Libor είδαμε και το θέμα κυρώσεων για νέες χειραγωγήσεις για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στην Ευρώπη και το σύνολο των χρηματοοικονομικών αγορών χρειαζόμαστε μια σαφή ρύθμιση που θα παρακολεί, θα αποκλείει η χειραγώγηση δικτών. Όχι μόνο την χειραγώγηση δικτών, αλλά να αποφύγουμε το να υπάρχουν κακοσχεδιασμένοι δείκτες, στρεβλοί δείκτες που θα δίνουν μια στρεβλή εικόνα που θα δίνει την δυνατότητα να δημιουργούνται φούσκες ή ανισορροπίες στις χρηματοοικονομικές αγορές. Η σοσιαλιστική ομάδα αξιολογεί θετικά αυτή την πρόταση ε, σε σχέση με την πρόταση που έχει υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να είμαι σύντομος θα επικεντρώσω την παρέμβασή μου σε τρία ή τέσσερα σημεία που πιστεύω ότι θα απαιτήσουν ένα πιο έντονο έργο, σε βάθος έργο κατά τις επόμενες εβδομάδες. Πρώτα απ' όλα, ο κανονισμός εκκινεί από έναν ορισμό κριτικού δίκτυ benchmarks, κριτικού χαρακτήρα, που θεωρώ μη ενδεδειγμένο αυτό το χαρακτήρα μια μέτρηση αποκλειστικά ποσοτική από την οποία απορρέει αν είναι κριτικός ή όχι, κρίσιμος ή όχι αυτός ο δείκτης. Νομίζω δημιουργείται εδώ, αφήνεται ένα κενό ε, ρυθμιστικό ε, και αυτό δεν είναι εύθετο. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να μετρηθούν και να αξιολογηθούν, να αποτιμηθούν ε, τα ε, κονδύλια ή πόροι και θα άφηνε ένα νομικό κενό για δείκτες που μπορούν ίσως να χρησιμοποιηθούν ε, με κέριο χαρακτήρα για την σταθερότητα των αγορών ή δείκτες που θα ήταν κέρι για την οικονομία κάποιων κρατών μελών αλλά που δεν είναι ίσως κέρια σημασίας για την Ευρωζώνη και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένας δίσκαμπτος αποκλειστικά ορισμός των κρίσιμων benchmarks. Πρώτον επειδή δημιουργείται ένα κενό ρυθμιστικό, ένα ενώ Δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος να σταθμιστούν και να αξιολογηθούν, να αξιολογηθούν τα κονδύλια που χρησιμοποιούν τέτοιους δείκτες. Και υπάρχει η δυνατότητα κάποιων δικτών που θα ήταν ασταθείς. Δεύτερο θέμα επί των οποίων έγινε αναφορά προηγούμενα είναι η αναλογικότητα, η αναλογικότητα της ρύθμισης. Είναι νομίζω ευκταίο να υπάρξει αναλογικότητα, λογική, εύλογη είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ισοπεδωτική ρύθμιση για το Γιούρι το του ή τους μεγαλύτερους δείκτες που έχουν ε, μεγαλύτερη δυνατότητα αποσταθεροποίησης των αγορών από ότι δείκτες που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς ή κλάδους αποκλειστικά ή σε περιφερειακές μόνο οικονομίες χωρίς συστημική α το πω έτσι επίπτωση. Πρέπει λοιπόν να θεωρείται η αναλογικότητα μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο. Να δούμε ποια είναι η λογική ε, που θα καθορίζει τους ε, κρίσιμους κέριους δίκτες και ποιους όχι. Και ένα τρίτο στοιχείο είναι το πρόβλημα της τρίτης χώρας, των τρίτων χωρών που σχολιάστηκε πιο πριν. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ελλειπής δεν υπάρχει τέτοια ρύθμιση και δεν μπορούμε να αφήσουμε εκτός ε, τις τρίτες χώρες, εκτός των benchmarks. Και τέλος, το πρότυπο εποπτείας ή επιτήρησης που πρέπει να καθοριστεί. Συγχαρητήρια και πάλι στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη η ε, κυρία Σουίνμπορν. Πολλά από τα θέματα τα οποία θέλω να δείξω έχουν καλυφθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την εισηγήτρια. Έγινε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τη εισηγήτρια και των σχεδόν εισηγητών και μπόρεσαν όλοι να εκφράσουν τι απόψει του στη διάρκεια τη διαδικασία. Οι τρει τομεί στους οποίου θα περιοριστώ είναι το πεδίο εφαρμογή, οι τρίτε χώρε και το διοικητικό άχθο. Καταρχά το πεδίο εφαρμογή. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο η ΑΙΟΣΚΟ έκανε δύο διαφορετικές εκθέσεις στον τομέα των δικτών αναφοράς. Η πρώτη έκθεση έγινε το 2012, όπου οι αρχές του ΑΙΟΣΚΟ για ε, όλους τις ε, ε, PRAs, τα γραφεία παρακολουθήσης των τιμών των βασικών προϊόντων και επίσης έγινε και μια διαφορετική έκθεση ε, για τελείως διαφορετικούς δείκτες αναφοράς. Έγιναν δύο διαφορετικές ε, εκθέσεις, διότι είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι που συγκεντρώνουν αυτούς τους δείκτες αναφοράς στους δύο τομείς. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές μεταξύ των χρηματοοικονομικών δικτών αναφοράς και αυτών που ετοιμάζουν τα γραφεία παρακολούθησης των τιμών των βασικών προϊόντων κυρίως για τις αγορές ε, αγαθών. Ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις διαφορές που υπάρχουν όπως για παράδειγμα τις ε, αγορές πετρελαίου και να αντιμετωπίσουμε και τις συγκεκριμένες δυναμικές κάποιων που συνεισφέρουν σε δείκτες αναφορές. Θα ήθελα να δω και όλους όσους συνεισφέρουν σε δείκτες αναφορές να συνεχίσουν να συνεισφέρουν σε περιοχέ όπω το Ιράν και η Ρωσία και να μην τους αποκλείσουμε ε, όταν θα είναι πολύ ψηλό ε, το άχθος για τα γραφεία παρακολούθησης των τιμών των βασικών προϊόντων για τα PRAs. Επομένως, ε, θεωρώ ότι το πεδίο εφαρμογής ε, για τους δείκτες αναφοράς πρέπει να είναι ξεχωριστό για αυτά τα προϊόντα από ότι για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Τώρα, στο διοικητικό άχθος. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι η βασική, η κρίσιμη ε, χρηματοοικονομικοί δείκτες αναφορές θα πρέπει ε, να λαμβάνονται δεόντως υπόψη και πρέπει να αποφασίσουμε όταν δεν είναι κρίσιμοι αυτοί οι δείκτες ε, να έχουν τελείως διαφορετικό καθεστώς από αυτούς που θεωρούνται κρίσιμοι. Και εδώ θα ήθελα να ζητήσω από όλα τα μέλη να δουν τι ακριβώς έγινε και στη χώρα μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον κανονισμό για τα Λίμπορ. Πλέον υπάρχει κανονισμός για πάνω από ένα χρόνο και είναι πολύ αυστηρές οι προδιαγραφές οι οποίες εφαρμόζονται όσους συνεισφέρουν και σε αυτούς που συγκεντρώνουν τους συγκεκριμένου δείκτες αναφορές. Αντί να επινοήσουμε εκ νέου κάτι καινούριο, καλό θα ήταν να δούμε τι κάνει ο κανονισμός Λίμπερ, διότι εφαρμόζεται και έχουμε νέους κανόνες αυτή τη στιγμή. Επίσης θα ήθελα να ε, πω εδώ ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την ποικιλομορφία για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτής της διατήρησης της ποικιλομορφίας, πρέπει να υπάρχουν διάφανε στοιχεία για τους δείκτες αναφορές, ώστε να λαμβάνονται καλές αποφάσεις για το ποιοι δείκτες αναφορές θα χρησιμοποιούνται, αλλά θα πρέπει να δούμε αν προσπαθούμε να επιβάλλουμε ε, σε όλους τους χρήστες ε, την ιδιότητα των αυτών που συγκεντρώνουν τους δείκτες. Εάν απλώς τροποποιείται ένας δείκτης αναφοράς, θεωρείται ότι είναι άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί δείκτη αναφοράς και είναι διαχειριστής του δείκτη, θα πρέπει να είναι σαφές λοιπόν αν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή σε δείκτη αναφοράς, ε, εάν περιλαμβάνονται σε αυτό το πεδίο ή όχι. Όσον αφορά τις τρίτες χώρες αναφέρθηκαν τα πράγματα, αλλά επειδή δεν υπάρχει πουθενά κάποια νομοθετική πρόταση στον κόσμο, θα πρέπει να προσέξουμε να μην επιβάλλουμε προδιαγραφές όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν θα μπορέσουν να τις στηρίσουν. Ε, θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο να βρούμε έναν τρόπο να εφαρμοστούν όταν θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένε αποφάσεις. Και αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Νίτερ ζητά να γίνει η αξιολόγηση επιπτώσεων ε, από το ερευνητικό τμήμα του Κοινοβουλίου. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα, θα ήθελα να το υποστηρίξω και εγώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη κι εγώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο διαθέσιμο για τη συνεδρίαση για αυτό το θέμα ούτως ή άλλως. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την παρουσίαση και τα σημεία που ανέφερε. Δυστυχώς σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους ε, δεν υπήρχε η ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτές τις συναντήσεις και αλλά μπορούμε να συνεργαστούμε, μπορούμε να δώσουμε συνέχεια. Γενικά συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έκανε η συγγήτρια. Για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν και από κάποιους από τους συναδέλφους επίσης χρειαζόμαστε σαφώς βελτίωση στον κανονισμό για τις ε, χρηματοπιστωτικές ε, benchmarks. Κάποιες από τις που έγιναν από την εισηγήτρια βαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση και είναι κέριος, κέρια σημασία σε αυτό το στοιχείο. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε είδους χειραγώγηση και τα άλλα πολλά προβλήματα παράλληλα τα οποία ούτως ή άλλως υφίστανται και αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους. Ως προς αυτό δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα προαναφέρθηκαν. Θέλω κάποια κέρια, κυριότερα στοιχεία να αναφέρω που θα ήθελα να ληφθούν υπόψη συζητώντας τα θέματα αυτού του χαρτοφυλακίου. Ένα από αυτά τα στοιχεία για μένα που είναι κέρια σημασίας είναι σχετίζεται με τις πτυχές που σχετίζονται με παραβιάσεις του δεοντολογικού κώδικα και δημιουργούνται συγκρούσεις συμφερόντων θα έπρεπε να υπάρχει ένα αυστηρότερο πλαίσιο και θα ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να εξετάσουμε. Δεύτερο, το εύρος. Πολλά πράγματα αναφέρθηκαν για το φάσμα, για το εύρος αυτών των μέτρων. Όμως το εύρος των benchmarks σε σχέση για παράδειγμα με την, τον υποχρεωτικό χαρακτήρα αυτών των στοιχείων θα μπορούσε να διαβρινθεί το εύρος τους και μπορούμε να το συζητήσουμε πιο εξειδικευμένα πρώτο σημείο για την ακαιρεότητα όσον αφορά την αξιοπιστία στην παραγωγή και εκπόνηση δικτών. Αυτό απαιτεί κάποια όρια να θεσπιστούν όσον αφορά τον εθελοντικό χαρακτήρα ροής αυτών των στοιχείων όσον αφορά τους διαχειριστές τους ώστε να είναι σαφέστερα τα πράγματα σε ένα σαφέστερο πλαίσιο. Ένα άλλο που θα ήθελα να αναφέρω ως παρατήρηση είναι η εφαρμογή, η υλοποίηση μεταβατικών προσωρινών ε, περιόδων όσον αφορά την αλλαγή μεθοδολογικής προσέγγισης. Πιστεύω ότι πρέπει να εισαχθεί αυτού του είδους ε, η μεταβατική περίοδος σε σχέση με τις αλλαγές που ε, σκοπεύουμε να εισαγάγουμε, όπου είναι δυνατόν να γίνει. Κατά αυτή την περίοδο τα benchmarks θα υπολογίζονται με βάση αρχές και της προηγούμενης αλλά και της νέας μεθοδολογίας σε μια τέτοια μεταβατική περίοδο λαμβάνοντας υπόψη διαφοροποιημένα την ε, ανάγκη χρήσης αυτών των στοιχείων και για τρίτες χώρες επίσης ε, που θα πρέπει να καλυφθεί και η πτυχή των τρίτων χωρών μπορούμε πιο εξειδικευμένα να το δούμε αυτό μελλοντικά ευχαριστώ ευχαριστώ για τους πράσινους εσείς έχετε τον λόγο παρακαλώ ευχαριστώ Όσον αφορά τις απογοητευτικές περιπτώσεις ε, χρηματοοικονομικών ε, σκανδάλων, σκανδάλων δείχνουν αυτά ότι η συμφωνία κυρίων ε, ήταν κάτι το οποίο δεν λειτουργούσε επαρκώς και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να υπάρξουν επαρκείς ρυθμίσεις ώστε να μπορούν τα πράγματα να λειτουργήσουν καλύτερα. Όσον αφορά τους μη αξιόπιστους δείκτες για παράδειγμα και τις, τις χειραγωγήσεις που υπήρξαν σχετικά είναι σαφές πλέον ότι πρέπει να διασφαλίσουμε εκπονώντας τέτοιου είδους προτάσεις ότι θα καλύπτονται όλες ε, οι ανάγκες, όλες οι πτυχές, γιατί για παράδειγμα όλες οι χειραγωγήσεις αντιβαίνουν την ορθή λειτουργία της αγοράς και είναι εις βάρος τους. Τα σκάνδαλα καταδεικνύουν, ότι πολλές φορές η νομοθεσία δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα επαρκώς. Αυτό τονίζει τη σπουδαιότητα να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και επιβολής και εποπτείας των benchmarks και να υπάρξει ένα ε, τέτοιο ισχυρό πλαίσιο το οποίο να αποβαίνει προς όφελος της Ευρώπης εισάγοντας στην ομοθεσία την αναλογικότητα και το εύθετο όμως ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μελλοντικά μπορούν όλα αυτά να επιτευθούν και να δικαιολογηθούν. Πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι σε σχέση με πολλά πράγματα υπάρχουν αμφισβητήσεις. Το να εισαχθούν λοιπόν νέες πτυχές που θα συμπεριλαμβάνουν τον ορισμό τέτοιων κινδύνων για να μπορέσουν να διαφοροποιηθούν σε σχέση με τους περιφερειακούς χαρακτήρα κινδύνους και αναφορά στη ρήτρα αναθεώρησης ότι θα πρέπει κατά την 1η Ιουλίου 2018 να δούμε την ανάγκη επανεξέτασης ε, αυτών των κανονισμών. Άλλες συγκεκριμένες προτάσεις θα διασφαλίσουν ότι όλα τα benchmarks νομοθετικά θα δημιουργούν ένα καθεστώς όπου θα ελέγχονται επαρκώς τα benchmarks για τις επιπτώσεις τους ε, και τους ε, κινδύνους που συνεπάγονται για το χρηματοοικονομικό σύστημα και θα ξέρουμε σε ποια ε, πλαίσια έχουν επιπτώσεις αυτά και θα θέλαμε να δώσουμε την δυνατότητα άμεσα να εξεταστούν τα κέρια σημασίας benchmarks. Να υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης τέτοιων προτάσεων μέσα στο πιο αποτελεσματικό πλαίσιο και να δούμε τις ε, τεχνικού χαρακτήρα προδιαγραφές που απαιτούνται ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και... Η Νίνα εκεί τώρα. Για το Καστιάι. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να πω ότι Ιστορικά τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματογορών και οι δείκτες αναφοράς προχωρούν χέρι-χέρι και σας εύχομαι καλύτερη τύχη από ό,τι σε μένα. Ε, απλώς να πω ότι χρειαζόμαστε μια συνολική λύση, κάτι πολιτικό, δεδομένου ότι έχουμε το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο ε, για την παραποίηση των τιμών και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο συνάδελφος, ότι δεν θα πρέπει να έχουμε μία αυστηρή ε, προσέγγιση και ένα αυστηρό καθεστώς απαραίτητος. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ποια είναι η αποψή σας όσον αφορά την εποπτεία. Ε, θέλετε να δώσετε περισσότερες εξουσίες στην ΕΣΜΑ ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι εθνικού χαρακτήρα η εποπτεία. Επομένως, έχω κάποια ερωτηματικά για τις εκκλήσεις για την αξιολόγηση επιπτώσεων, γιατί το θέμα αυτό έχει εξεταστεί εδώ και αρκετό καιρό και πραγματικά δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να πετύχουμε αν είχαμε μια νέα αξιολόγηση επιπτώσεων. Εγώ πραγματικά σας κούρω τον κόδωνα του κινδύνου ε, από αυτού. Ευχαριστώ η Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιοδείς συζητητές και την κυρία Γκίλ φυσικά για τις απόψεις της και τις απόψεις όλων των υπολείπων. Νομίζω ότι μας περιμένει σκληρή δουλειά τις επόμενες εβδομάδες, αλλά ε, την περιμένουμε ανυπομονησία αυτή τη δουλειά, γιατί βλέπω ότι όλοι έχουν αυτή την αίσθηση του κατεπήγοντος. Πρέπει να είναι πιο αυστηρός ο κανονισμός και κάτι πρέπει να γίνει από αυτού. Εάν λοιπόν όλοι ε, τραβάμε προς την ίδια κατεύθυνση τη διελκυστίδα, νομίζω ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Όσον αφορά την αξιολόγηση επιπτώσεων, εγώ αν κατάλαβα καλά, ο κ. Νίτερ Μάιερ δεν ζήτησε να υπάρχει μια νέα αξιολόγηση επιπτώσεων θέλει απλώς και μια δεύτερη γνώμη για την αξιολόγηση επιπτώσεων που έχει ήδη ε, συνταχθεί, ε, που αφορά κυρίως τις τρίτες χώρες και τα προβλήματα των χωρών αυτών. Δεν ζήτησε λοιπόν μια νέα ε, αξιολόγηση επιπτώσεων, εξ όσων γνωρίζω εγώ, αν κατάλαβα καλά. Ε, βλέπω κάποιους άλλους και να γνέφουν καταφατικά, οπότε μάλλον αυτό ζήτησε. Και λαμβάνοντας και πάλι υπόψη το γεγονός ότι θεωρούμε όλοι ότι πρέπει επιγόντως να κάνουμε κάτι, ε, δεν νομίζω ότι θα καθυστερήσει τα πράγματα, αλλά ο κύριος Νίτρη Μαέμ μας είπε ότι δεν θα έπρεπε να καθυστερήσουν λογικά και ελπίζω να ισχύει αυτό που μου είπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμίες τώρα. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης 8 Ιανουαρίου, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 20 Ιανουαρίου, εξέταση στις 23 Ιανουαρίου, ψηφοφορία 5 Μαρτίου. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο θα ξεκινήσουμε στις 8 το πρωί σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Επασχόλησης. Έχουμε πλέον ε, αίθουσα. Μου είπαν ότι θα υποθέτω ότι είναι γνωστό. Εδώ στην αίθουσα λοιπόν.